Ξεκινάμε την ε, συνεδρίαση την πρακτική ε, της, συνεδρία, της ε, Επιτροπής μας μετά από την κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση για τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω τον συνάδελφο Βίλαν, τον αντιπρόεδρο, που έχει γίνει μέλος αναπληρωματικό της Επιτροπής μας. Σας χαιρετίζουμε λοιπόν με χαρά διότι οι νομικές σας γνώσεις σίγουρα θα λύσουν πολλά προβλήματα, ε, κυρίως ρυθμιστικού χαρακτήρα. Κατά τα λοιπά, ήδη εργάζεται σε μια ομάδα ad hoc που θα χρειαστεί να παρακολουθήσει και να μας δώσει δείξη, υποδείξη μεθόδους για να παρακολουθήσουμε τη συμμετοχή των βουλευτών σε μεγάλες σημαντικές στιγμές συζήτησης του Κοινοβουλίου, πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε κάθε ποιες προτάσεις για ε, τροποποίησης του κανονισμού. Μέγα κύρος λοιπόν προσδίδει στη σημερινή συνεδρίαση όπως και του συναδέλφου Πέτερινγκ η συμμετοχή. Ε, πολύ σημαντικός ο ρόλος του και συναδέλφου Βίλαντ. Ορισμένες ανακοινώσεις όσον αφορά τις συνεδρίες των συντονιστών χτες ώστε να μπορέσετε να τις επικυρώσετε τις προτάσεις Στη Βουδαπέστη 9 και 10 Δεκεμβρίου 2010 θα γίνει μια συνάντηση μιας δικής μας αντιπροσωπείας με εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου και του ακαδημαϊκού κόσμου καθώς και της κοινωνίας των πολιτών της Ουγγαρίας. Η αντιπροσωπεία θα πρέπει να αποτελείται λοιπόν από μένα για το ΕΛΚ, Ταρκόφσκι, Λεγκρίπ και Σέρπνιγκ ο οποίος είναι εκτός κότα επειδή είναι Ούγγρος. Αυτή τη φορά λοιπόν είναι έξι οι συμμετέχοντες. Για τους ε, σοσιαλιστές θα είναι ο κύριος Γκερέρο και η κυρία Γκουρμά που είναι και εκείνη εκτός ε, ποσόστοση. Άλντε Νταφ και Πράσινη Έφνερ και ο κύριος Σόλτς ε, επίσης. Και αν όλοι συμφωνείτε αυτοί θα είναι οι συμμετέχοντες. Άλλη την προσωπία θα πάει στο Κέμπριτζ 27-28 Ιανουαρίου 2011 να προετοιμαστεί καλύτερα η ε, επίσκεψη. Θα το συζητήσουμε αργότερα για το ποιοι θα συμμετέχουν. Οι συντονιστές εξέτασαν επίσης την ε, ανταπόκριση σε αιτήματα βουλευτών εθνικών κοινοβουλίων άλλων κρατών που θέλουν να έρθουν ε, σε συνάντηση με δική μας αντιπροσωπεία. Είπαμε να είμαστε αρκετά ευέλικτοι, να υποδεικνύουμε κατά προτίμηση τις ημέρες όπου ε, συνεδριάζει η Επιτροπή μας, ώστε οι αντιπροσωπείε των άλλων χωρών να μπορούν να συμμετέχουν στι εργασίε μα, αλλά αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, να είναι εγγυημένη μια συνάντηση σε επίπεδο προεδρίας ή, ή κάποιας εκπροσώπησης προεδρίας. Νομίζω πως Μιλήσαμε και για ένα προσανατολισμό άλλο, να ζητήσουμε δηλαδή από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ την δυνατότητα να υποβάλουμε γνωμοδότηση για την ε, έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ σε σχέση με την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας και όσον αφορά τη δικασία απαλλαγή προπολογισμού για το 2009, οι συντονιστέ θεωρούν πω δεν χρειάζεται εμεί ω Επιτροπή να συντάξουμε γνωμοδότηση. Αυτές είναι οι ανακοινώσει από δική μου πλευρά. Δεν βλέπω παράτηρήσει από τη δική σας πλευρά, άρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην εξέταση μερίσιας διάταξη που προβλέπει το σημείο 8 τη. 8 που εν μέρη ήδη Εξετάστηκε η μερίσια διάταξη και το 8 αφορά την εφαρμογή του κανονισμού 2004-2003 σχετικά με το καθεστώ και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπω ξέρετε, αυτό ο κανονισμό προβλέπει μέχρι το Φεβρουάριο του 2011 το Κοινοβούλιο να εγκρίνει μια ανέκθεση για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Στην πράξη, μα ανετέθη εμά ω την ΑΦΚΟ να υποβάλουμε έκθεση για το θέμα και η συγκεκριά μα ήδη έχει οριστεί από τις 18 Οκτωβρίου είναι η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. το Προεδρείο του Κοινοβουλίου έχει γκρίνει μία πρόταση για την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και περιμένει από εμάς τη γνωμοδότηση, την έκθεσή μας. Δεν μου μένει τίποτα άλλο να κάνω, να δώσω μόνο το λόγο στην συνάδελφο Γιαννάκου που νομίζω θα μας υποδείξει τα βασικά στοιχεία της παρέμβασης αυτής ε, της έκθεσής μας και θα μας πει και για χρονοδιάγραμμα για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πράγματι όπως ε, αναφέρατε και εσείς θα πρέπει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου να υπάρξει ε, η έκθεση αυτή του Κοινοβουλίου η οποία βασίζεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του κυρίου Βέλεμ προκειμένου σχετικά με την αξιολόγηση της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Πρέπει ευθύ αμέσω να σας πω ότι η έκθεση του κυρίου Βέλε έγινε εγκαίρος από το μήνα Σεπτέμβριο. Το Προεδρείο όμως άργησε πάρα πολύ ε, να εγκρίνει στη συνεδρίασή του την έκθεση αυτή με αποτέλεσμα το όριο της 15ης ε, Φεβρουαρίου να μην είναι εφικτό. Δηλαδή θα ήθελα λίγο να σας μιλήσω για το χρονοδιάγραμμα. Όπως ακριβώς ε, συνεννοηθήκαμε και συζητήσαμε με τη Γραμματεία. Καταρχήν προτείνεται να γίνει μια δημόσια ακρόαση ειδικών τον μήνα Ιανουάριο. Και γιατί προτείνεται, ε, γιατί υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον για το ζήτημα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων αφενός και για το καθεστώς των πολιτικών κομμάτων, όπως ακριβώς εδώ αναφέρεται στον τίτλο ε, και έτσι έχουμε συζητήσει με τη γραμματεία και βέβαια είναι αποδεκτές και οι προτάσεις των συντονιστών και των διαφόρων πολιτικών ομάδων ε, να γίνει ένα hearing στις 26 Ιανουαρίου από ειδικού, είτε στα θέματα διαφάνειας, είτε στα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν, είτε στα οικονομικά. Να παρουσιαστεί το πρώτο σχέδιο έκθεσης πέντε μέρες μετά, στις 31 Ιανουαρίου του 2011 η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών να είναι η 17η Δευτέρου 2011, να υιοθετηθεί στην Επιτροπή στις 15 Τρίτου 2011, 15 Μαρτίου και στην Ολομέλεια να μπει τον Απρίλιο. Ε, το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μπορεί να υιοθετηθεί καθώς και την προηγούμενη φορά το 2006 που είχε γίνει η έκθεση αξιολόγησης με βάση τον κανονισμό του 2003 επίσης είχε εγκριθεί το Μάρτιο η έκθεση. Επομένως νομίζω ότι προτείνω δηλαδή να αποδεχθούμε αυτή τη μικρή καθυστέρηση που δεν οφείλεται σε εμά πάντως ούτε και στο Γενικό Γραμματέα. Το πρόγραμμα της ακρόασης βέβαια νομίζω θα συζητηθεί, δεν χρειάζεται να σας το αναλύσω αυτή τη στιγμή. Ε, θέλω να σημειώσω ε, ότι η πρόταση κανονισμού έτσι όπως τροποποιήθηκε το 2007, δηλαδή η πρόταση του 2003, έχει οδηγήσει σε ένα πιο ευέλικτο και λιγότερο γραφειοκρατικό σύστημα χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών κομμάτων και κατά την εκτίμηση που έχω κάνει Νομίζω ότι ικανοποιεί τα περισσότερα κόμματα με τους γενικούς γραμματείς των οποίων βέβαια εγώ θα συζητήσω σε σχέση με την έκθεση του κυρίου Βέλε και προφανώς θα κληθούν στην ακρόαση ε, να εκφράσουν την άποψή τους. Ε, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία ε, στην προσεχή έκθεση είναι αυτό που πολλές φορές έχει συζητηθεί εδώ στο Κοινοβούλιο ε, για την ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού κανονισμού που να διέπει και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων μια που υπάρχει αντίστοιχη τέτοια χρηματοδότηση. Ε, επομένως ε, είναι ζήτημα που αφορά στην έκθεση αξιολόγησης για το ποια διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού κοινού καθεστώτος για τη δημιουργία και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Ε, νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι είναι άλλωστε κάτι το θέμα αυτό ε, το οποίο ε, θα μπορούσε, μπορεί να έχει και δημοσιότητα εν συνεχεία διότι όπως γνωρίζετε και σε εθνικό επίπεδο πολλές αμφισβητήσεις υπάρχουν σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις των κομμάτων και κατά καιρού δημιουργούνται διάφορα θέματα. Εμείς λοιπόν νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, να παρουσιάσουμε με τον πιο διαφανή και καθαρό τρόπο ε, την χρηματοδότηση αυτή και την πεποίθηση που μπορεί να δημιουργηθεί στον κόσμο ότι εν πάση περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί όλους τους σχετικούς κανόνες και τις αρχές διαφάνειας που πρέπει να διέπουν μια τέτοια χρηματοδότηση. Σε μια εποχή άλλωστε γενικότερης οικονομικής κρίσης κύριε Πρόεδρε, παρακολουθώντας και τον τύπο και το διεθνή τύπο αλλά και στη χώρα μου, ε, βρίσκω πολλά σχόλια τα οποία τις περισσότερες φορές δεν είναι και πραγματικά ούτε σωστά ε, σχετικά με το κόστος της Ευρώπης, ιδιαίτερα από ορισμένε πολιτικές πλευρές αν θέλετε, και νομίζω ότι ε, με την έκθεση αυτή θα απαντήσουμε και πολύ καθαρά ε, για το ποια είναι η σκοπιμότητα και η ωφέλεια ε, από την χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κομμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Γιαννάκου. Η γνωμοδότηση αυτή, η έκθεση αυτή μάλλον είναι πολύ σημαντική, γιατί δεν αφορά μόνο το οικονομικό θέμα, είναι και πολιτικό. Είναι ένα ζήτημα επίκαιρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία χρειάζεται τα πολιτικά κόμματα. Και με τον συνάδελφο Νταφ μιλούσαμε για, μια ομοιόμορφο, για έναν ομοιόμορφο εκλογικό νόμο. Φυσικά ένας ε, νόμος εκλογικό σε λειτουργεί όταν υπάρχουν και πολιτικά κόμματα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των πολιτικών κομμάτων. Θέλει κανεί το λόγο από τα μέλη τη Επιτροπή, ο κύριο Νταφ. Συμφωνώ ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό κύριε Πρόεδρε και θα πρέπει να το χειριστούμε κατάλληλα και να του δώσουμε τη δέουσα προσοχή. Θα ήθελα να εξετάσουμε το σημείωμα του Κλάους Βέλε, του Γενικού Γραμματέου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την εφαρμογή του δημοσιονομικού κανονισμού. Μήπως θα μπορούσατε λοιπόν να μας μοιράσετε αυτό το σημείωμα του Γενικού Γραμματέα, ήταν πολύ χρήσιμο. Ε, έμαθα ότι το Ρεπουμπλικάνικο κόμμα στις πρόσφατες ε, ενδιάμεσες ε, εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες δαπάνησε 4 δισεκατομμύρια δολάρια 4 δισεκατομμύρια δολάρια, επαναλαμβάνω, στην προεκλογική του εκστρατεία. Οπότε, όταν αντιμετωπίζουμε τις επικρίσεις του σκεπτικιστικού τμήματος του τύπου για την διεύρυνση των οικονομικών διευκολύσεων για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, δεν χρειάζεται να είμαστε και πολύ αμυντικοί όταν έχουμε τέτοια παραδείγματα αλλού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκερέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά τη γνώμη μου, η έκθεση αυτή και ο κανονισμός είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε χωρίς κανένα αίσθημα ενοχής, κανένα απολύτως αίσθημα ενοχής, αλλά θα πρέπει να προασπίσουμε τα ουσιώδη στοιχεία και αυτό που βρίσκεται πίσω από το θέμα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Και ως σκιώδης συγκητής των σοσιαλιστών θα ήθελα καταρχήν να δηλώσω ότι τα πολιτικά κόμματα σε πολλά από τα συντάγματα των χωρών μας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της κοινή γνώμης και επίσης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην έκφραση της λαϊκής βούλησης. Πρόκειται για σημαντικούς θεσμούς λοιπόν για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας. Και στην περίπτωση Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πολιτικά κόμματα είναι σημαντικοί θεσμοί για την ίδια την ευρωπαϊκή οικοδόμηση και ολοκλήρωση και για την, ε, με τους, την ε, εσάρκωση της ηθαγένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την έκφραση της βούλησης των πολιτών για τη μελλοντική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι θεσμικός και συνταγματικό ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων και πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό και η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, όποια και είναι η μορφή που τελικά θα επιλέξουμε, η χρηματοδότηση αυτή είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του συστήματος. Μάλιστα, αν κάνουμε μια σύγκριση των εμπειριών μας, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν διάφορες μορφές χρηματοδότησης. Σε ορισμένες χώρες έχουμε ιδιωτική χρηματοδότηση κατά κανόνα. Σε άλλες κρατική χρηματοδότηση και σε ορισμένες χώρες ένα μείγμα ιδιωτικής και κρατικής χρηματοδότησης. Όλος παραδόξως, η ιδιωτική χρηματοδότηση εχμαλωτίζει πολύ περισσότερο τα πολιτικά κόμματα από τη δημόσια χρηματοδότηση. Η ιδιωτική χρηματοδότηση προκαλεί πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση των πολιτικών κομμάτων από την ε, χρηματοδότηση του κράτους. Γι' αυτό, χωρίς κανένα κόμπλεξ και χωρίς καμία ενοχή, εμείς θα πρέπει να διεκδικήσουμε δημόσια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Πολιτικών Κομμάτων. Τώρα, η αντιστοιχία σχέση με αυτά που προτείνουμε είναι να θεσπίσουμε ένα κανονισμό που θα εξασφαλίζει σαφήνεια σε ό,τι αφορά του τρόπου χρηματοδότηση. Η σαφήνεια για τη χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντική. Επίση, η διαφάνεια είναι πολύ σημαντική για τα τμήματα αυτής της χρηματοδότησης και φυσικά λογοδοσία των πολιτικών κομμάτων για τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, δεν θα πρέπει να είμαστε αμυντικοί, να εθετήσουμε αμυντική θέση, γιατί τα πολιτικά κόμματα έχουν θεμελιώδη ρόλο τη λειτουργία ενός δημοκρατικού συστήματος. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να επιλέξουμε μια δημόσια χρηματοδότηση γιατί εξασφαλίζει καλύτερα την ανεξαρτησία των πολιτικών κομμάτων και επίσης θα πρέπει να συνοδεύσουμε αυτή τη δημόσια ε, χρηματοδότηση με σαφήνεια, διαφάνεια και λογοδοσία. Και νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να είναι τα βασικά στοιχεία του κανονισμού που θα εγκρίνουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κεραίρο. Τρεις ε, συνάδελφοι έχουν ακόμη ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Βίλαντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια όταν με υποδεχθήκατε. Το θέμα του κόστους που έδειξε ο κύριος Ντάφ. Είναι περιορισμένος ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επικαλεστούμε την κατάσταση στην Αμερική. Όταν μιλούμε για τα 4 δισεκατομμύρια, τα χρήματα αυτά προέρχονται κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα και από μικρούς και από μεγάλους, αλλά λιγότερο μεγάλους. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε σύγκριση με το κόστος αυτό. Πρέπει να θέσουμε το ερώτημα, θέλετε τέτοιου είδους δημοκρατία όπου υπάρχουν τέτοιες ενδεχόμενες εξαρτήσεις στο θέμα του κόστους θα ήθελα να τονίσω και οι δύο κύριοι της Γραμματείας γνωρίζουν καλά την κατάσταση, σχετικά με το καθεστώς των Ευρωβουλευτών δηλαδή, ήδη από την εποχή Ρότλαϊ είχαμε κάνει και συγκρίσεις αριθμητικών στοιχείων. Τι στοιχίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία να διατηρηθούν και να συνεχιστούν να τηρούνται, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προέκυπτε από αυτά, παρόλο το μεγάλο κόστος των γλωσσικών εργασιών και των τριών εδρών εργασίας κατά κεφαλήν κοστίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λιγότερο από τα νομοθετικά όργανα των ΗΠΑ, κατά κεφαλήν δηλαδή Ευρωπαίου πολίτη. Όπως ε, νομίζω θα πει και ο κ. Λαμπρινίδης, σε ένα σημαντικό θέμα της εκθέσης αυτής θα είναι από πότε αρχίζει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κόμμα. Χρειαζόμαστε ας πούμε πέντε ευρωβουλευτές. Χρειαζόμαστε ας πούμε συμμετοχή οκτώ χωρών όπου να έχει κάποιο ποσοστό το συγκεκριμένο κόμμα έστω και αν δεν υπάρχουν Ευρωβουλευτές Χρειάζονται για παράδειγμα τρεις βουλευτές Για παράδειγμα, στη Βάδη Βιρτεμβέργη, αν, κάποιος έχει, αν κάποιο κόμμα έχει τρει βουλευτέ, μπορεί να πει ότι είναι Ευρωπαϊκό Κόμμα. Άρα μέχρι να γίνει ακρόαση θα πρέπει να ψάξουμε, να μελετήσουμε και συγκριτικά στις χώρες μας δηλαδή, να δούμε από ποια στιγμή αρχίζει στο εθνικό δίκαιο των χωρών μελών, έτσι, να χαίρει κάποιων νομικών προνομίων ένα κόμμα, να συμμετέχει σε εκλογές, ποια πρέπει να είναι η δύναμη ενός κόμματος στις χώρες μέλη ώστε να μπορεί να μπει σε πιο νομικό επίπεδο, ώστε να έχει όχι μόνο οικονομικά προνόμια, αλλά και νομικά. Για παράδειγμα, αλλάζουν συχνά οι πρόεδροι των κομμάτων. Εάν κανείς έχει ένα σωματείο στην Γερμανία και αλλάζει πρόεδρο, αυτός πρέπει να εγγραφεί στο αρχείο του ειρηνοδικίου. Ενώ τα κόμματα δεν έχουν την υποχρέωση αυτή Λοιπόν, από ποια αριθμητική δύναμη και μετά, ως κόμμα, ποια προνόμια αποκτά το συγκεκριμένο κόμμα, λοιπόν, από ποια αριθμητική δύναμη και πάνω, στις χώρες μέλη. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε και συγκριτικά, λοιπόν. Και όποιος θέλει να γνωρίζει κάτι για την Ευρώπη θα έχει πολλά να πληροφορηθεί από αυτά. Και παρακαλώ την εισηγήτρια να σκεφτεί εάν ίσως θέλουμε, από, και από, θέλουμε στην ακρόαση να συμμετάσχει και κάποιος από το ελεγκτικό συνέδριο. Διότι η διαμόρφωση των οικονομικών θα έχει σχέση και τι γίνεται και με τους μέχρι τώρα δημοσιονομικούς κανονισμούς των θεσμικών οργάνων. Δύο παραδείγματα είναι προκειμένου. Το Νοέμβριο του 2010, εφόσον είμαι εγώ ας πούμε πρόεδρος κόμματος και σχεδιάζω το τι πρωτοβουλίες θα αναλάβω το 2011. Δεν μπορώ να ξέρω, ας πούμε, για τον Αύγουστο του 2011 τι θα ήθελα να κάνω. Θέλω να κάνω πέντε workshop, πέντε εργαστήρια, θέλω να κάνω μια μεγάλη διάσκεψη. Όμως, ο δημοσιονομικός κανονισμός προβλέπει και απαιτεί ακριβή ε, διαμόρφωση των σχεδιασμών αυτών Εάν δεν κάνουμε κάποιες αλλαγές εδώ, δεν μπορούμε λοιπόν να ανταποκριθούμε στις υποχρώσεις αυτές. Δεύτερο, ακούστηκε κάτι περί δημιουργικότητας. Α, με συγχωρείτε, όχι. Ευκαμψία, ευελιξία. Αν έχουμε υπερβολική ευκαμψία, υπάρχει και ένας κίνδυνος δημιουργικότητας εντός εισαγωγικών. Άρα να παραμείνουμε στο μέσον της οδού, να δούμε πού ακριβώς χρειάζονται αλλαγές, πού πρέπει να διατηρηθούν κάποια πράγματα. Άρα η γνώμη μου και η συμβουλή μου είναι να ζητήσουμε οδηγίες, να ζητήσουμε συμβουλές από ανθρώπους του ελεγκτικού συνεδρίου, να δούμε δηλαδή ποια πράγματα είναι δυνατόν να γίνουν και εκεί όπου θα μας πει το ελεγκτικό συνέδριο προσοχή αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν, να δούμε ποιες αλλαγές πρέπει να προκύψουν στον δημοσιονομικό κανονισμό. domanda, eh, suo intervento l'ha fatto ad una... Ε, αναφερθήκατε σε μια ανάγκη τεκμηρίωσης, πράγμα που ήδη συμβαίνει. Διερωτώ με όμως αν υπάρχει όμω ένα είδο έκθεση όσον αφορά τον τρόπο χρηματοδότηση των κομμάτων στα μεμονωμένα κράτη-μέλη, στα εκάστοτε κράτη-μέλη. σω η Κομισιόν να έχει ήδη κάνει κάποια τέτοια μελέτη. Ε, Θα ήταν σκόπιμο λοιπόν και γι' αυτό, αυτό να απασχολεί στην ακρόαση. Ο κύριος Μπρόνς. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε η βασική μου θέση είναι ότι είμαι κατά της εθνική κρατικής χρηματοδότησης, τη ε, κοινοτική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Ε, παίρνουν ε, πόρους από τα μέλη τους και από τους υποστηρικτές τους. Και αν όχι, αυτό συμβαίνει λόγω έλλειψης σοβαρότητας. Οι επίσης μπορεί να χρηματοδοτούνται από επιχειρήσει ή συνδικάτα ή σωματεία. Κατά την άποψή μου ούτε αυτό θα πρέπει να επιτρέπεται γιατί τα κόμματα τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από τέτοιους πόρους θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Θα πρέπει, λοιπόν, αν, λοιπόν τελικά επιτραπεί χρηματοδότηση από την κοινότητα, θα πρέπει αυτό να υπόκειται σε αντικειμενικά και συγκεκριμένα κριτήρια. Δεν μπορεί να αλλάζει με στόχο να ευνοήσει κάποια κόμματα και να μειώσει κάποια άλλα, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν ιδιαίτερα μετά από τις, ε, την τροπολογία Κόρμπετ το 2009. Ορισμένοι λένε σήμερα το πρωί πω τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι ζωτική σημασία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει αφοσίωση σε ένα ευρωπαϊκό κείμενο ολοκλήρωση πριν να, μάλλον να βρεθεί συμφωνία για χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κομμάτων. Μάλιστα, σα ευχαριστώ. Ο κύριο Λαμπρινίδη. <clears throat> Um, Επιτρέψτε μου να θίξω λίγα από τα κυριότερα στοιχεία της εκθέσεως του Γενικού Γραμματέως όπως συζητήθηκαν αυτά στην διάρκεια του τελευταίου Προεδρίου και να σας μεταφέρω την έννοια των συζητήσεων αυτών και ορισμένες προσωπικές απόψεις. Ένα από τα πιο κύρια σημεία, όπως είπε ο κύριος Βίλαντ και άλλοι, είναι το πώς θα ιδρύεται, το πώς θα δημιουργείται το Ευρωπαϊκό Κόμμα. Ένα κόμμα το οποίο να μπορεί να δεχθεί και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Στη διάρκεια των συζητήσεων στο Προεδρείο διαφάνηκε μεγάλη πλειοψηφία και ελπίζω να εξεταστεί και από την παρούσα Επιτροπή ότι τουλάχιστον ένας ευρωβουλευτής θα είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται, να υπάρχει δηλαδή από το κόμμα αυτό ώστε να μπορεί να λάβει αυτό ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Όπως έχουν οι κανονισμοί σήμερα, φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα να ιδρυθούν ευρωπαϊκά κόμματα και να λάβουν και σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έστω και αν έχουν μόνο κάποιους περιφερειακούς εκπροσώπους σε κάποιες χώρες, χωρίς καμία νομιμοποίηση στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα δεύτερο θέμα ήταν η νομική προσωπικότητα του Ευρωπαϊκού Κόμματος. Εκεί διεξήχθη μεγάλη συζήτηση και όχι εύκολη. Ζητήσαμε από την Γραμματεία να συντάξει ένα σύντομο σημείωμα μελέτη σχετικά με αυτό που ο κ. Βίλαντ σχετικά δηλαδή, δηλαδή με τις αρχικές προϋποθέσεις στις διάφορες χώρες μέλη αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου που να είναι συμβατά με τις δικές μας εδώ ε, υποθέσεις ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με το ποιο θα πρέπει να είναι το νομικό πλαίσιο. Φαίνεται ότι η πλειοψηφία θεωρεί ότι είναι ελλειπές το παρόν νομικό πλαίσιο, αλλά πώς θα πρέπει να συμπληρωθεί και αυτό δεν είναι απόλυτα σαφές. Η συζήτηση ελπίζω ότι θα συμβάλλει στην διευκρίνηση του θέματος αυτού. Τώρα, άλλο θέμα που συζητήσαμε και είναι από τα κύρια σημεία της εκθέσεως του σημειώματος δηλαδή του Γενικού Γραμματέως είναι τα ευρωπαϊκά ιδρύματα, η δυνατότητα δημιουργίας αποθεματικών. Το Προεδρείο φαίνεται να έχει τη γνώμη ότι κάτι τέτοιο θα ήταν σωστό, αλλά δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Έχουμε κάνει μια αρχική συζήτηση μόνο και τίποτα περισσότερο. Επίσης θα πρέπει να, υπάρχει, να υπάρξει ένα ειδικό ταμείο για τις ευρωεκλογές, μάλλον για τις ευρωπαϊκές προεκλογικές εκστρατείες. Μία πρόταση λέει ναι, μία άλλη πρόταση λέει να υπάρχει μια αύξηση στη διάρκεια του έτους των εκλογών των προϋπολογισμών των κομμάτων αναλογικά με την δύναμή τους και με αυτά που λαμβάνουν για να διεξαγάγουν προεκλογικές εκστρατείες. Αυτό πάντως είναι αίτημα όλων των κομμάτων και είναι εύλογο. Ένα θέμα που ακούστηκε σήμερα εδώ έχει σχέση με τις δωρεές. Συμφωνώ με τον κύριο Γκερέρο σχετικά με τη σημασία της δημόσιας χρηματοδότησης. Αυτό είναι σαφές. Οι κανονισμοί των ευρωπαϊκών κομμάτων σήμερα προβλέπουν και ιδιωτικές δωρές και προβλέπουν και μια οροφή για τις δωρές αυτές. Το, το Προεδρείο συζήτησε αν θα πρέπει να αυξηθεί η οροφή ή να παραμείνει ή και αν αυξηθεί για κατά πόσον. Ο Γενικός Γραμματέας προτείνει μια αύξηση που κατά τη γνώμη μου είναι υπερβολικά υψηλή. από ένα όριο 10 έως 12.000 που είναι οροφή σήμερα, φτάνει μέχρι 50.000 ο Γενικός Γραμματέας ανά ιδιωτική δωρεά. Εμένα αυτό μου φαίνεται υπερβολικά υψηλό. Θα το συζητήσουμε βέβαια στο Προεδρείο, θα συζητήσουμε ποιες εναλλακτικές επιλογές υπάρχουν, αλλά αφού διαλαμβάνεται στην πρόταση του Γενικού Γραμματέως, θα πρέπει να το συζητήσει το θέμα αυτό και η παρούσα Επιτροπή. Γενικά, Πάντως κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε στο Προεδρείο ότι το έργο που έχει κάνει η γραμματεία του Προεδρείου είναι εξαιρετική, είναι εντελεχής και μάλιστα για ένα θέμα πολύ περίπλοκο. Εγώ σας τόνισα ορισμένα από τα θέματα που συζητήσαμε, ίσως το, τα πλέον επίμαχα αν θέλετε, ασφαλώς υπάρχουν και άλλα. Πάντως γενικά η αίσθηση που έχουμε είναι ότι κινούμαστε στην σωστή κατεύθυνση με τις συστάσεις αυτές. Τα πολιτικά κόμματα με τα οποία συζητήσαμε και ο κύριος Βίλαντ και εγώ φαίνεται να συμφωνούν και σε ό,τι αφορά την διαφάνεια ας πω το εξή. Εμείς πιστεύουμε και συστήνουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ελεγκτής ένα όργανο ελεκτικό το ίδιο για όλα τα πολιτικά κόμματα που θα χρηματοδοτείται από εμάς που θα ελέγχει όλα τα κόμματα στην Ευρώπη με τα ίδια κριτήρια και είναι νομίζω εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει αυτή η βεβαιότητα ότι τα ίδια δηλαδή κριτήρια εφαρμόζονται από τους ίδιους ανθρώπους που θα έχουν επιλεγεί αντικειμενικά. Θα εφαρμόζονται λοιπόν σε όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα είναι πραγματικά ένα βήμα αποφασιστικής σημασίας προς την προς μια μεγαλύτερη διαφάνεια. Ασφαλώ και θεωρώ ότι τα ευρωπαϊκά κόμματα είναι σημαντικά, πρέπει να υποστηριχθούν, αλλά πρέπει να γίνει υποστήριξη αυτή με διαφάνεια. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κανεί άλλο το λόγο. Μόνο η συγκήτρια, η κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε σημείωσα όσα ελέγχθησαν. Θέλω να σας πω καταρχήν ότι ήδη προβλέπεται ότι το ελεκτικό συνέδριο θα συμμετάσχει στην ακρόαση. Θα συμμετέχουν επίσης καθηγητές εγνωσμένου κύρους οι οποίοι έχουν γνώση σχετικά με τα καθεστώτα των κομμάτων και του συνταγματικού δικαίου καθηγητές οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν την ε, γνώση τους γύρω από τα θέματα Τρίτον, θα συμμετάσχει, θα προσκαλέσουμε τη διεθνή διαφάνεια. Ε, να μας πει την άποψή της γενικότερα, όχι για τη συγκεκριμένη έκθεση βέβαια και την αξιολόγησή της ε, και για τα συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία, ε, αλλά γενικότερα για το στατή των ευρωπαϊκών κομμάτων και τι θα σήμαινε βέβαια ε, ένα τέτοιο καθεστώς και η προς τα έξω κοινοποίηση ε, και της χρηματοδότησης ε, των πολιτικών, ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων που πρέπει να είναι δημόσια. Όπως γνωρίζετε βέβαια τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ήδη χρηματοδοτούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρηματοδοτούνται βέβαια και από τα κόμματα μέλη τους τα οποία συμβάλλουν σε κάτι τέτοιο και αμφιβάλλω αν υπάρχει ουσιαστική χρηματοδότηση η οποία γίνεται από διάφορους δωρητές. Στην ακρόαση επομένως θα κληθούν οι γενικοί γραμματείς όλων των κομμάτων με τους οποίους άλλωστε θα συζητήσω και εγώ πολύ πριν ε, από την ακρόαση αυτή προκειμένου να εκφράσουν την άποψή τους και να μιλήσουν και για τα αντίστοιχα ιδρύματα, για τα, φοντα... για τα foundations τα οποία υπόκεινται και υπάγονται στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Επομένως η συζήτηση και η διαβούλευση με όλους αυτούς όσους ε, ε, εμπλέκονται ασφαλώς είναι δεδομένη και ασφαλώς από πλευρά εισηγητού θέλω να σας βεβαιώσω ε, ότι φυσικά είμαι υπέρ μιας ε, αυστηρής και απαρέγκλητης εφαρμογής ε, των όποιων κανονισμών προκρίνονται η αναφορά μου στην ευελιξία είναι γιατί αναφέρεται πραγματικά και στην έκθεση ε, του Γενικού Γραμματέα και βέβαια σας υπενθυμίζω ότι ο κανονισμός του 2003 τροποποιήθηκε το 2007. Δηλαδή αφού είχε γίνει η προηγουμένη έκθεση αξιολόγησης η οποία γίνεται ανά ε, το 2006. Επομένως κύριε Πρόεδρε αν η Επιτροπή εγκρίνει αυτό το χρονοδιάγραμμα ε, ενδιαμέσως και ως ότου γίνει το hearing ε, θα υπάρξει ένα πρώτο σημείωμα εν συνεχεία και αφού έχουν γίνει συζητήσεις με όλους όσους σας ανέφερα θα γίνει η ακρόαση αυτή η έκθεση ώστε να καταλήξουμε εν καιρό να εγκριθεί τον Απρίλιο από το Κοινοβούλιο. Αυτό που έχει πολιτική σημασία, το οποίο αντιλαμβανόμεθα όλοι, είναι η έννοια του καθεστώτος ε, ενός Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος, διότι πράγματι κύριε Πρόεδρε, και εγώ συμφωνώ ότι τα κόμματα αποτελούν παράγοντες της δημοκρατίας και επομένως το καθεστώς και οι κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία τους ε, έχουν σχέση με την ε, ε, άμεση τήρηση των κανόνων της δημοκρατίας και σε εθνικό αν θέλετε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως η αξία, η συζήτηση αυτή γίνεται υπό το φως υποθέτω ε, της αναγνώρισης από όλους μας της αξίας των πολιτικών κομμάτων ε, και ως θεσμικών παραγόντων και ως πρακτικών μέσων για να μπορεί να εκφραστεί λαϊκή βούληση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το θέμα αυτό. Από πλευρά τη Επιτροπή μα, ε, θεωρώ πω ε, ε, συμφωνείτε με το προθεσμίε που μα εξέθεσε η κυρία Γιαννάκου. 26 Ιανουαρίου και 31 θα γίνει συζήτηση. Γενικά είναι ευνοϊκή, ευνοϊκός ο προσανατολισμός όσον αφορά τη σημασία του θέματος, τόσο όσον αφορά τη χρηματοδότηση των κομμάτων, που ε, θα είναι μάλλον δημόσια, κρατική, και αναγνωρίζεται η ανάγκη για μια, ένα καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων που να είναι ξεκάθαρο συνεπές και να μπορεί να προωθήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ευχαριστούμε κυρία Γιαννάκου και προχωράμε στο επόμενο σημείο της της διάταξης που αφορά την πρωτοβουλία πολιτών. Είναι το τελευταίο θέμα για σήμερα. Όπως γνωρίζετε, Ήδη έχουν ε, δουλέψει εντατικά, έχουμε συζητήσει το έγγραφο εργασία, έχουμε κάνει μια πρώτη γενική ακρόαση με εκπροσώπου των Εθνικών Κοινοβουλίων, μια δεύτερη ακρόαση πιο συγκεκριμένα με ε, πυρογνώμονε για το θέμα και σήμερα θα πρέπει να παρουσιαστεί από τους συζητητέ την κυρία Γκουρμάη και τον κύριο Λαμασούρ το σχέδιο έκθεσης μετά από αυτό δε ε, πρέπει να αναθέσουμε υπό το σύμφωνο με το άρθρο 70 εντολή ώστε να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσει με τη, ε, άλλα θεσμικά όργανα. Υπάρχουν ε, πολλές σημαντικές προοπτικές, υπάρχει ταυτότητα απόψεων πάνω στα βασικά σημεία, οπότε ευχόμαστε ε, ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ταχύτατη και οριστική έγκριση στην πρώτη ανάγνωση. Αυτό σημαίνει όμως ότι επισήμω θα πρέπει να δώσουμε εντολή σε μια κάποια δική μας αντιπροσωπεία. Δίνω το λόγο στους εισηγητές. Ε, νομίζω ότι έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων να μιλήσει η κυρία Γκουρμάη. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ αλλά όπως ξέρετε είναι κοινό το έργο, άλλη φορά αρχίζει ο Αλέ, άλλη φορά αρχίζω εγώ, αυτή τη φορά έχω την τύχη να αρχίζω εγώ. Πάντως είναι κοινή η προσπάθεια και ευχαριστώ θερμά όχι μόνο τον Αλέ αλλά και όλους τους συναδέλφους γιατί χάρη στην πολύτιμη συνεισφορά όλων καταφέραμε και συνεργαστήκαμε πολύ θετικά. Όλοι γνωρίζουμε ότι η πρωτοβουλία των πολιτών είναι ένα θέμα πολύ επίκαιρο σε όλες τις ευρωπαϊκές συζητήσεις μετά την πολύ ε, σφοδρή συζήτηση που είχαμε και την εκστρατεία για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών είναι μια μοναδική ευκαιρία για να δώσουμε νέα πνοή ζωής στην ευρωπαϊκή δημοκρατία και να ενισχύσουμε την συμμετοχή των πολιτών στην ε, διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχύσουμε τη συζήτηση για, τις, για τα διάφορα ευρωπαϊκά θέματα. Το άρθρο 11, παράγραφος 4 της Συνθήκης Λισαβόνας, δεν λέει και πολλά πράγματα. Λέει ότι ε, ένα εκατομμύριο υπογραφές ε, Ευρωπαίων πολιτών χρειάζονται για να αναλυφθεί πρωτοβουλία και να προσκληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της να υποβάλει οποιαδήποτε πρόταση για θέματα για τα οποία οι πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική δράση της Ένωσης προκειμένου να εφαρμοστούν οι συνθήκες. Τώρα εναπόκειται σε εμά, τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, να βρούμε με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει αυτή η διάταξη στην πράξη. Η Επιτροπή Αναφορών, μάλιστα, ε, συζήτησε αυτό το θέμα και γι' αυτό ο Ζεράρ και η Νταϊάννα, οι συνεισηγητές, θα έρθουν αργότερα, ε, όπως και πολλοί πρόσωποι του Συμβουλίου. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε πλήρη επίγνωση των ευθυνών μας και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στις τελευταίες ευρωεκλογέ μόνο 42% των Ευρωπαίων πολιτών προσήλθαν στις κάλπες. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την ε, θέσπιση αυτού του νέου οργάνου. Και αν ε, θέλουμε νομοθεσία που θα προβλέπει ασφαλή και αποτελεσματική χρήση, θα γεφυρώσουμε αυτό το περίφημο χάσμα μεταξύ μόν και των συμπολιτών μας. Βέβαια υπάρχουν υψηλές προσδοκίες ε, για την πρωτοβουλία αυτή των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει να αποφύγουμε την απογοήτευση και ματέωση αυτών των προσδοκιών. Γιατί ήδη είδαμε ότι άρχισε η συγκέντρωση υπογραφών ε, για διάφορα θέματα. Βέβαια θα πρέπει να πούμε στους πολίτες ότι δυστυχώς παρά την ε, άοκνη προσπάθειά μας δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη την διαδικασία αυτή. Το σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υπευλήθη το Μάρτιο είναι μια πολύ καλή πρόταση και σημείο αφετηρία. Ήρθε, ήρθαν και ο Μάριο και η Γκάμπριελ από το επιτελείο του Μάρος Σεφτσοβιτς, του Αρμοδίου Επιτρόπου, και οι συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχθηκαν ότι χρειάστηκε να τηρήσουν ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα κατά την εκπόνηση του εγγράφου. Ελπίζω πάντως ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι διαλλακτική ε, και απέναντι στις δικές μας προτάσεις. Με βάση τον κανόνα 50, όπως είπα, η Επιτροπή Αναφορών έχει ήδη ξεκινήσει τη συζήτηση και είχαμε πολύ αγαστή συνεργασία και με την Ισπανική Προεδρία. Μάλιστα, έχουμε εκπονήσει και ένα έγγραφο εργασία ε, στα πλαίσια της Ισπανικής Προεδρίας. Πήραμε πολύ στα σοβαρά το έργο μας και η Ισπανική, Ουγγρική και Βελγική Προεδρία, το τρίο ε, φυσικά ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Είχαμε πολύ θετική συνεργασία και με τη Βελγική Προεδρία και θα ήθελα να θα ευχαριστήσω θερμά τον Ελβια Σαστέλ και το επιτελείο του. Θα δούμε αν και η επόμενη Ουγγρική Προεδρία συνεργαστεί το ίδιο θερμά μαζί μας. Είχαμε πολυάριθμες συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη για το θέμα της πρωτοβουλίας των πολιτών, όχι μόνο με βουλευτές αλλά και με εκπροσώπους κρατών μελών. Και όπως είπε και ο Πρόεδρος, είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε και με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή Περιφερειών δραστηριοποιήθηκαν για το θέμα αυτό. Και ο ε, ε, ε, εξέφρασε τη γνώμη του για αυτό το νέο εργαλείο, το νέο μηχανισμό το νέο τέκνο κατά κάποιο τρόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο δημιούργημα, για μας ε, τα πράγματα είναι απλά. Θέλουμε όσο δυνατόν περισσότερες πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων πολιτών. Θέλουμε πραγματικά οι Ευρωπαίοι πολίτες να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία και γι' αυτό χρειάζονται πολλές αλλαγές, είναι απαραίτητες πολλές αλλαγές στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να είναι πρακτικό και εύχριστο αυτό το εργαλείο της πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων πολιτών. Μία τέτοια πρωτοβουλία θα ευοδοθεί φυσικά αν ο κανονισμός είναι φιλικός προς τον χρήστη, προς τον πολίτη και δεν δημιουργεί φοβερές γραφειοκρατικές διατυπώσεις και γραφειοκρατικό άχθο για τους συμμετέχοντες. Αυτό είναι λοιπόν ο στόχος μας, να βελτιώσουμε το σχέδιο του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπή προκειμένου να γίνει πιο φιλικό προ τον χρήστη. Σε χαιρέτησα και πριν Μάριο, αλλά μια και ήρθε στο λέω και διαζώσει. Θέλουμε περισσότερε πληροφορίε για την πρωτοβουλία αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να είναι ένα ισχυρό δημοκρατικό εργαλείο να μην γίνει κατάχρησή του, να είναι αποτελεσματικό για του πολίτε και να το αξιοποιούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν ο μηχανισμό αυτό να είναι ένα εργαλείο τη συμμετοχική δημοκρατία που θα είναι προσιτό προ ευρωπαίου πολίτε και θα αφορά ευρωπαϊκά ζητήματα. Αυτό χρειαζόμαστε και φυσικά θα πρέπει η διαδικασία να γίνει όσο πιο ευρωπαϊκή γίνεται ευθύ εξ αρχή και να ε, διευκολυνθεί η διασυνοριακή διακρατική συνεργασία και η διακρατική συζήτηση. Έχουμε 7 συναδέλφους από 7 διαφορετικές ε, χώρες μέλη, οπότε ε, δημιουργούνται οι για μια πανευρωπαϊκή συζήτηση. Φυσικά μερικές φορές ε, το, η προϋπόθεση της ε, απέτηση ενός ελάχιστου αριθμού υπογραφών από συγκεκριμένο κρατος είναι υπερβολικά γραφειοκρατική. Δεν θα πρέπει να προσκρούσουμε στο δύσκολο εγχείρημα της συγκέντρωσης ενός εκατομμύριου υπογραφών. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα. Πώς είναι δυνατόν ε, να, συγκεντρωθούν τα μέσα για τη συγκέντρωση τόσων υπογραφών. Η η Επιτροπή των Πολιτών λοιπόν θα πρέπει να διευκολυνθούν και να αντιμετωπίσουν λιγότερες δυσκολίες για τη συγκέντρωση των υπογραφών που απαιτούνται. Ακόμη και από την ε, αρχή υπάρχει το δίκτυο των ε, εκπροσώπων στα ενδιαφερόμενα κράτη που περιμένουν για την επίσημη, την επίσημη πράξη έναρξη της συγκέντρωση των υπογραφών. Επίσης θέλουμε όσο πιο πολλές ε, μεταφράσεις γίνεται. Εγώ προέρχομαι από μια μεσαία χώρα σε μέγεθος και η ουγγρική γλώσσα είναι καταπληκτική, θέλουμε την ευκαιρία να το αποδείξουμε. Επίσης, ε, η πληθώρα πολιτών από πολλές χώρες θα διευκολύνει τις περισσότερες μεταφράσεις. Βέβαια, αυτό ίσως δημιουργεί ένα πρόβλημα για την Επιτροπή των Πολιτών, γιατί η μετάφραση είναι λίγο γραφειοκρατική. Γι' αυτό και η Επιτροπή προτείνει, δύο βήματα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του παραδεκτού. Πώς θα εξηγήσουμε στους ε, πολίτες ότι μπορούν να ξεκινήσουν μια πρωτοβουλία, μπορούν ε, να, να συγκεντρώσει 300.000 υπογραφέ, μετά θα πρέπει να περιμένουν δύο μήνε ώστε να εξεταστεί το παραδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανάλογα με το τι θα αποφασίσει να δουν αν θα μπορούσαν να συνεχίσουν ή όχι. Σαν να είναι χαμένο όλο ο κόπο δηλαδή αυτό που έκαναν. Δεν θα πρέπει να ζητούμε από του ε, πολιτε να ε, υπογράφουν μια πρωτοβουλία που ίσω κριθεί μη παραδεκτή. Αυτό είναι μια ματαιοπονία. Ελπίζω τελικά να καταλήξουμε σε συμφωνία για το σημείο αυτό. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι και η πρωτοβουλία αυτή, όπω κάθε δικαίωμα, συνοδεύεται από πολλέ υποχρεώσεις και διοικητικέ που προσπαθούμε να τις ελαχιστοποιήσουμε, αλλά και σεβασμό των ε, θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, μεταξύ άλλων ε, προϋποθέσεων. Επίσης, ε, θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη διατύπωση, γι' αυτό και περιλαμβάνουμε μνήα του άρθρου 2 τη συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ευθυγράμμιση τη διαδικασία με τις απαιτήσει προστασία δεδομένων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης να εξασφαλίσουμε απόλυτη διαφάνεια τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος της. Οποιοδήποτε κόμμα σωματείο μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια πρωτοβουλία πολιτών αρκεί να υπάρχει πλήρης διαφάνεια ώστε να ξέρουμε ποιο βρίσκεται πίσω από μια πρωτοβουλία και να το γνωρίζουν αυτό οι πολίτε για να επιλέξουν αν θα υποστηρίξουν την πρωτοβουλία ή όχι. Η έκβαση των πρωτοβουλειών θα είναι κέρια σημασία και θα πρέπει η έκβαση μιας πρωτοβουλίας να αντικατοπτρίζει το έργο και των οργανωτών θα πρέπει και η Επιτροπή να εξηγεί τις δράσεις που θα στηρίζονται στην πρωτοβουλία και να αιτιολογεί την απόρριψη σε περίπτωση που δεν συμφωνήσει να δώσει συνέχεια σε μια πρωτοβουλία. Θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το μονοπόλιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας, αλλά θα πρέπει να είναι σαφής απέναντι στους πολίτες. Επίσης, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν την εξασφάλιση ότι θα γίνει και μια δημόσια κρόση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συνεργάζονται προκειμένου να οργανώνουν τέτοιου είδου συζήτηση για μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Και όλα αυτά θα πρέπει να είναι γνωστά και διαφανή. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτε να έχουν σαφή και εξαντλητική ενημέρωση για το πώς λειτουργεί ή μια πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών για όλους τους τομείς, από τα κριτήρια ε, καταχώρησης μέχρι την τελική δημόσια κρόση, καθώς και πιθανά μέσα προσφυγής. Θα πρέπει να υπάρχει ένα help desk από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό αποδείχθηκε από τις ε, τελευταίες συζητήσεις. Περιμένουμε και τα σχόλιά σας γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει σύσσωμο να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία με νέο μέτωπο, αν θέλουμε πραγματικά αυτός ο νέος μηχανισμός να είναι επωφελής για τους συμπολίτε μας και νομίζω ότι όλοι αισθανιζόμαστε αυτό το στόχο. Θέλουμε η πρωτοβουλία των πολιτών να γίνει μια λειτουργική και εύρυθμη πραγματικότητα, γιατί το χρωστάμε αυτό στου πολίτε μα. Ήδη έχει περάσει ένα χρόνο από τη θέση ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα και εύλογα θα διαρωτώ οι πολίτε γιατί να μην μπορούμε ακόμη να χρησιμοποιήσουμε αυτό το νέο δημοκρατικό μηχανισμό. Εγώ μπορώ να πω ότι εργαζόμαστε άοκνα προκειμένου ο μηχανισμό αυτό να τεθεί στη διάθεση των πολιτών το συντομότερο δυνατό. Θα πρέπει όμω όλοι να γνωρίζουν ότι η πίεση χρόνου θα πρέπει να αποβεί βάρο τη ποιότητα του έργου μα. Και ω ε, ε, υπεύθυνοι πολιτικοί και βουλευτέ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε σωστή χρήση της πρωτοβουλίας αυτής προκειμένου να ικανοποιεί τους συμπολίτες μας. Μάλιστα εδώ μπαίνουμε σε μη χαρτογραφημένο έδαφος, για, σε μια πρωτοφανή και άνευ προηγουμένου ρύθμιση. Είναι σαν να πηδάμε σε μια λίμνη, να βουδάμε σε μια λίμνη που δεν ξέρουμε πόσο βαθιά και πόσο μεγάλη είναι. Γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επιτυχή εφαρμογή του μηχανισμού και να μην ξεχνούμε ότι στην πορεία μπορεί να ανακύψουν πολλά θέματα που ούτε τα διανόμαστε τώρα. Γι' αυτό και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει έκθεση εφαρμογής ε, τακτική για την εφαρμογή του κανονισμού και δεχομένω να προτείνει και αναθεώρηση του κανονισμού σε περίπτωση που κρυθεί απαραίτητο. Ευχαριστώ, αλλά σε λίγο θα έρθουν και τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών, φαντάζομαι. Ελπίζω να τα καταφέρουμε, γίνεται στην πρώτη ανάγνωση και ελπίζω να συνεργαστούμε όλοι προς αυτόν τον σκοπό. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκορμάη για αυτήν την ε, ενδελεχή έκθεση. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Λαμασούρ που είναι ο συνεισηγητής. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά και Συμφωνώ με τα όσα είπε η Αντιπρόεδρος Γκουρμάη και χαίρομαι για την ποιότητα των σχέσεών μας κατά την εκπόνηση αυτού του κοινού, της κοινής έκθεσης. Εγώ θέλω μόνο να συμπληρώσω δύο λόγια για κάποια σχόλια για τη μέθοδο εργασίας και για το περιεχόμενο. Για την μέθοδο, από την πρώτη μέρα κιόλα, εμείς εκφράσαμε την επιθυμία εντός του Κοινοβουλίου μαζί με τα άλλα θεσμικά όργανα, τα ευρωπαϊκά, αλλά και εκτός, να δουλέψουμε με τελείως ανοιχτό τρόπο και μέσα σε ένα μόνιμο διάλογο, με την βούληση να φτάσουμε σε όσο γίνεται ευρύτερη συμφωνία. Και συγκεκριμένα στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο να έχουμε όσο γίνεται πιο μεγάλη πλειοψηφία. Καθώς ε, δεν θέλουμε να φτιάξουμε μια διαδικασία δεν θέλουμε να έχουμε, δεν, δεν είναι ιδιωτελής η επιλογή, αλλά θέλουμε να φτιάξουμε μια διαδικασία ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μια πολύ καινοτόμα διάταξη της συνθήκης της Λισαβόνας που ενδιαφέρει τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Όχι μόνο λοιπόν χάρη στην ε, σοφία σας, αλλά και χάρη, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής ε, ε, Συνταγματικών Υποθέσεων, και συνθέσαμε μια ομάδα τεσσάρων εισηγητών, δύο συνεισηγητών στο πλαίσιο της ΑΦΚΟ, ώστε οι τέσσερις κέρυες ομάδες να αντιπροσωπεύονται στην ομάδα που θα προετοιμάσει το σχέδιο έκθεσης. Διάφορες επιτροπές του Κοινοβουλίου θα υποβάλουν γνωμοδοτήσεις και πολλοί από τους εισηγητές των γνωμοδοτήσεων είναι εδώ για να συμμετέχουν στη συζήτηση αυτή και έχουμε τόσο στο πλαίσιο της Επιτροπής ΑΦΚΟ όσο και στο πλαίσιο των πολιτικών ομάδων αλλά και σε άλλα πλαίσια προέβημεν σε διάφορες ακροάσεις και ανταλλαγέ απόψεων συμπεριλαμβανομένες της δικής σα προεδρίας κύριε Πρόεδρε με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και ως πολιτικό στόχο θέσαμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα που θα μας επιτρέψει την υιοθέτηση του κανονισμού σε μια μόνο ανάγνωση το Δεκέμβριο. Και είχαμε και διάφορες άτυπες επαφές, έπειτα πιο επίσημες επαφές, χωρίς να έχουμε εντολή συντονιστή βέβαια από το στάδιο. Συγγνώμη. Φυσικά μπορούν και να μας απαλλάξουν αν δεν θεωρούν πως δεν ε, ακολουθούμε το σωστό δρόμο. Για το περιεχόμενο, φιλοσοφία μας είναι να εφαρμόσουμε ολόκληρη τη συνθήκη. Όλα όσα επιτρέπει η συνθήκη. Και με πρώτη προτεραιότητα τους πολίτες, δηλαδή να είναι όλα αυτά φιλικά προς τον πολίτη. Αυτό μα οδήγησε σε διαφορετικές, ε, σε μάλλον προτεραιότητες σε σχέση με τα όσα μας, αρχικά μας πρότεινε η Κομισιόν. Ποιο είναι ο στόχο τη συνθήκης. Ο στόχο της συνθήκης είναι να δώσει στους πολίτες μια δυνατότητα να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι η ίδια με αυτή που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω των ψηφισμάτων που εγκρίνει και με αυτήν που έχει τη δυνατότητα το Συμβούλιο. Δηλαδή από εδώ και μπρος τρεις κατηγορίες φορέων υπάρχουν. Το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και οι πολίτες που μπορούν να καλέσουν την Επιτροπή να δράσει. Ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Και άρα η ιδέα μας είναι να βρούμε τον τρόπο ώστε η διαδικασίες που θα δημιουργηθούν είναι εύκολες, απλές, προσβάσιμες για τους πολίτες. Για να μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν αυτό, αυτή τη δυνατότητα, όπως το εκμεταλλεύεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ένα δικαίωμα πρωτοβουλίας, δεν είναι συμμετοχή στην νομοθετική εξουσία. Είναι ένα δικαίωμα πολιτικής πρωτοβουλίας. Αλλά η νομική πρωτοβουλία παραμένει μονοπόλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό το μονοπόλιο σημαίνει, το θυμίζω, είναι η εξουσία αποκλειστική της Κομισιόν και αφορά την απόφαση για το αν είναι πολιτικό σκόπεμο να συνταχθεί νομοθετικό κείμενο. Αυτή η απόφαση ανήκει στην Κομισιόν, είναι το δικό της προνόμιο, και το μονοπόλιο και αν αποφασίσει πω χρειάζεται νομοθετικό κείμενο, φυσικά εκείνη συντάσσει και το σχέδιο. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο νομικά έχουν το δικαίωμα να εργαστούν πάνω σε κείμενα τα οποία καταθέτουν, καταθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θυμίζω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για να καταλάβουμε κάποιες από τις ε, συγκεκριμένες προτάσεις που κάνουμε. Όπως σας είπα, πρέπει να είναι ε, φιλικό προς τον πολίτη όσο γίνεται περισσότερο. Δικαιώματα του πολίτη, ναι, δικαίωμα στην απλοποίηση και εκεί κάναμε ένα γιγάντιο άλμα σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν που στην ουσία θα εμπόδιζε κάθε ε, κατάληξη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας ε, των πολιτών. Απέτηση δηλαδή 500 υπογραφών, το Συμβούλιο μίλησε για 100.000 και ξέρω εγώ. Πάση περιπτώσει, μη ρεαλιστικά πράγματα. Η πρόταση ήταν λοιπόν να σύγχωνε η, δυνατότητα καταγραφής και το παραδεκτό, ε, θέτοντας ως προϋπόθεση την συλλογή 7, 8, 9 υπογραφών που συγκεντρώνονται μέσα σε ένα πλαίσιο μια οργάνωση ανθρώπων που είναι συντάκτες της πρωτοβουλίας που θα πρέπει να έρχονται από ε, αντίστοιχα αριθμό χωρών και θα πρέπει να δίνουν και ένα συγκεκριμένο αριθμό εγγύησεων. Από τη στιγμή όμως που ξεκινά αυτή η πρωτοβουλία από ανθρώπους που προέρχονται από τον αριθμό των χωρών μελών που αντιστοιχούν στο μήνυμο που απαιτείται για να αναγνωρίζεται ως έγκυρη αυτή η πρωτοβουλία δεν υπάρχει άλλος όρος. Δεν υπάρχει ο άλλος όρος για να προτείνουμε για αυτές τις διατάξεις που σχετίζονται με την ε, πρωτοβουλία, ορισμένοι από του συζητητέ ε, για γνωμοδότηση δεν έχουν ακριβώ την ίδια άποψη όπω εμεί, α πούμε, για τη διάρκεια συλλογή των υπογραφών, αν είναι 12 μήνε, 18 μήνε ή κάτι άλλο. Για να διευκολύνουμε τα πράγματα, προσπαθήσαμε να επιτρέψουμε στους ε, ε, αρχικούς συλλέκτους των υπογραφών να συλλέξουν ένα συγκεκριμένο αριθμό υπογραφών με μήνυμο ηλικία νόμιμη ηλικία 16, ε, τα 16 έτη και δεν θα έχουμε δυσκολίες με το Συμβούλιο και προτείναμε ο αριθμός των χωρών να είναι το 1 πέμπτο, ενώ το Συμβούλιο και η Κομισιόν προτείνει το 1 τρίτο. Ταυτόχρονα για τα δικαιώματα των πολιτών δικαίωμα ενημέρωσης για την ίδια τη διαδικασία και για την κατάληξή της. Να εξηγηθώ τώρα. Δεν πρέπει να αφήνουμε τους πολίτες να δεσμευθούν σε μια διαδικασία αν δεν γνωρίζουν τις πιθανές, την πιθανή κατάληξή της ή μπορεί να ίσχυε κάποια παρεξήγηση και μια, μάλιστα μια προφανής παρεξήγηση που θα πρέπει να ε, εξαλειφθεί εξ αρχής και αυτό προτείνουμε να κάνουμε στην αιτιολογική έκθεση αλλά που θα πρέπει επίσης να το παρουσιάσουμε σωστά από τη στιγμή που θα αρχίσει να ισχύει ο κανονισμός. Δεν σημαίνει επειδή ένα εκατομμύριο υπογραφές συγκεντρώθηκαν ότι θα υπάρξει ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όχι. Είναι μια, μια δυνατότητα πολιτικής πρωτοβουλία, αλλά όχι νομοθετική εξουσία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική διάκριση. Δικαίωμα των πολιτών, δικαιώματα των πολιτών, αλλά και υποχρεώσεις από την άλλη των πολιτών. Α, όχι, συγγνώμη. Υπάρχει και ένα τελευταίο δικαίωμα που είναι επίση πολύ σημαντικό, που είναι το δικαίωμα σε μια πολιτική παρακολούθηση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η κατάληξη της ε, πρωτοβουλίας των πολιτών που θα πληρεί τους όρους κτλ δεν θα γίνεται συστηματικά, δεν θα είναι μάλλον μια νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία ή τροποποίηση τη ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό θα εξαρτηθεί από την εκτίμηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο για του πολίτε που θα υπογράψουν. Αντιθέτω, και επ' αυτού οι φίλοι τη Επιτροπή Αναφορών επέμειναν και συμφωνούμε σε αυτό και το έχουμε συμπεριλάβει στο σχέδιο έκθεση και μπορούμε και να το βελτιώσουμε. Αν λοιπόν συγκεντρωθούν ένα εκατομμύριο υπογραφέ, αυτοί οι πολίτες έχουν δικαίωμα για μια πολιτική παρακολούθηση, δηλαδή να γίνουν ακουστοί, να συζητηθεί το θέμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το εξετάσει και στην ε, περίπτωση που δεν δώσει νομοθετική συνέχεια, να εξηγήσει γιατί δεν δίνει νομοθετική συνέχεια και αν διαπιστωθεί ότι η ανησυχία των πολιτών είναι θεμητή αλλά ότι δεν ε, χρειάζεται να γίνει σχετική νομοθεσία έχουμε ηθική και πολιτική υποχρέωση να προσπαθήσουμε να δώσουμε άλλου είδους απαντήσεις σε αυτό το νόμιμο, την νόμιμη ανησυχία των πολιτών. Δικαίωμα των πολιτών λοιπόν απλή διαδικασία, πλήρη ενημέρωση για την ίδια τη διαδικασία και την κατάληξή της, τι επιτρέπει δηλαδή και τι όχι και εν πάση περιπτώσει, αν πάει μέχρι τέλο έχουν δικαίωμα για μια πολιτική ε, συνοδεία ή παρακολουθησία. Σε αντίβαρο υπάρχουν ε, κάποιες υποχρεώσεις. Ένα, ε, συντήρηση της συνθήκης και των αρχών αυτής. Αυτό είναι θεμελιώδες. Δεν ε, θέλουμε να εισαχθεί στον κανονισμό μια διάταξη που θα ξεπερνούσε τη συνθήκη. Αυτό δεν μπορεί παρά, η πρωτοβουλία μάλλον, να αφορά παρά μόνο ένα θέμα που είναι αρμοδιότητα της Ένωσης και για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταθέσει νομικό, νομοθετικό κείμενο. Άρα λοιπόν, τροποποίηση της συνθήκης ή σε σχέση με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράδειγμα δεν είναι αποδεκτές τέτοιες πρωτοβουλίες. Το μέσα στο αυτής της Το ίδιο ισχύει και για το σεβασμό των αρχών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, επίση άλλη απέτηση σημαντική είναι η διαφάνεια. Το συζητήσαμε επί μακρόν. Ξέρω ότι οι ορισμένες επιτροπές που γνωμοδοτούν έχουν διαφορετική άποψη σε σχέση με εμά και ενδιαφέρονται να συνεχιστεί η συζήτηση από κοινού σήμερα. Θεωρούμε λοιπόν πως αρκεί 8-9-10 πολίτες να υπογράψουν ένα σχέδιο πρωτοβουλία των πολιτών αν ανήκουν σε διαφορετικές χώρες και αυτό αρκεί για να ξεκινήσει να λειτουργεί ο μηχανισμό. Όμω έχουν την υποχρέωση να είναι απόλυτα διαφανεί όσον αφορά την πολιτική του στήριξη και την οικονομική του στήριξη. Μπορεί να το στηρίζει μια πολυεθνική, μπορεί να το στηρίζει ένα πολιτικό κόμμα, μπορεί να το στηρίζει πολιτικά και οικονομικά οποιοδήποτε. Ωραία, εντάξει, δεν απαγορεύεται, αλλά υπάρχει απόλυτη υποχρέωση διαφάνειας ώστε να ξέρουμε. Και να μην ψεύδονται σε αυτούς που θα ζητήσουν μετά τις υπογραφές. Τώρα, θέλαμε όπως σας είπα να είμαστε φιλικοί προς τους χρήστες αλλά και προς τα κράτη. Και θέλουμε να είμαστε φιλικοί προς τι κυβερνήσει, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανησυχίε τους. Οι ανησυχίες τους εστιάζονται στη δεύτερη φάση της διαδικασία, δηλαδή τη φάση συλλογή των υπογραφών και στην επαλήθευση των υπογραφών. Η πρώτη φάση είναι η καταγραφή. Καταγραφή και αποδοχή. Μετά ε, δεύτερη φάση είναι η συλλογή και τρίτη φάση είναι η πολιτική συνέχεια που δίνεται. Για τη δεύτερη φάση έχουμε μια βασική δυσκολία που είναι σημαντική γιατί εμείς θα θέλαμε και νομίζω πως είναι μια άποψη που είναι κοινή για όλες τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές δηλαδή να Έχουμε όσο γίνεται απλούστερο τρόπο για συλλογή των υπογραφών, ώστε να μην αποτρέπονται, αποτρέπονται πολίτες στους οποίους μπορεί να ζητάμε πολλά έγγραφα, διευκρινήσεις, πληροφορίες για την ταυτότητά τους και τα λοιπά, αλλά ταυτόχρονα από την πλευρά των κρατών μελών, στους οποίους θα βαραίνει ο έλεγχος της ταυτότητας των πολιτών, ο έλεγχος δηλαδή του ότι δεν υπάρχει διπλή υπογραφή και ότι οι άνθρωποι ε, όντω ε, που υπογράφουν είναι Ευρωπαίοι πολίτες, είναι άνω των 18 ή 16 ετών κτλ. κτλ. Άρα λοιπόν τα κράτη-μέλη χρειάζονται κάποιες εγγυήσεις. Μεγάλη δυσκολία είναι λοιπόν πως αυτές οι εγγυήσεις είναι τελείως διαφορετικές από κράτος σε κράτος. Και εδώ έχουμε πραγματικό πολιτικό πρόβλημα ουσίας ε, ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε αυτή τη φάση. Θέλουμε επίσης να είμαστε και φιλικοί προς την Κομισιόν φυσικά, αλλά εδώ νομίζω δουλεύουμε αρμονικά με την Κομισιόν και από τη στιγμή που ο καθένας σέβεται το ρόλο του, σύμφωνα με τις συνθήκες, θα βρεθεί αποδεκτή λύση για όλους. Θέλουμε επίσης να είναι φιλικό για το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα που τίθεται λοιπόν είναι από τη στιγμή που θα φτιαχτεί ο κανονισμός. Το ίδιο το κοινοβούλιο τι θα κάνει. Και αυτό θα πρέπει να το ε, μας απασχολήσει για να δούμε αν θα προβλέψουμε κάτι στον κανονισμό από τώρα. Για την ώρα η στάση μας είναι μάλλον περιοριστική. Δηλαδή, όσο λιγότερο γίνεται λόγος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτόν τον κανονισμό, τόσο περισσότερο θα μπορεί να ενεργήσει το Κοινοβούλιο και εξηγούμε. Δηλαδή, το Κοινοβούλιο μπορεί να ασχοληθεί με οποιοδήποτε θέμα μέσω μια έκθεση πρωτοβουλία ανα πάσα στιγμή. Κάθε μια από τι επιτροπέ μα μπορεί να αποφασίσει για μια δημόσια κρόαση ανα πάσα στιγμή. Και άρα εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία. Αν μια επιτροπή του Κοινοβουλίου, η Ολομέλεια ή μια πολιτική ομάδα του Κοινοβουλίου επιθυμεί να ενθαρρύνει μια πρωτοβουλία των πολιτών που είναι στην αρχή ή να ενθαρρύνει τη συλλογή πρωτοβουλειών ή αντίθετα να προειδοποιήσει κατά ορισμένων πρωτοβουλίων και θέλει να διοργανώσει συζήτηση πριν να ξεκινήσει ή να ολοκληρωθεί η συλλογή των, των υπογραφών, σήμερα τίποτα δεν το εμποδίζει. Αν το Κοινοβούλιο θέλει να παρέμβει από τη στιγμή που έχει συγκεντρωθεί ο αριθμός του 1 εκατομμυρίου υπογραφών και πριν να ενεργήσει η Κομισιόν, πάλι μπορεί να το κάνει. Ούτως ή άλλως επισήμως από την Κομισιόν θα έρθει έτοιμα από τη στιγμή που θα ε, ε, έχει γίνει αποδεκτό το αίτημα της πρωτοβουλία των πολιτών. Ακόμα και αν δεν μας προτείνει η νομοθετική διαδικασία θα είναι υποχρεωμένη να μας εξηγήσει γιατί κατά την αποψή της η ανησυχία των πολιτών δεν χρειάζεται να οδηγήσει σε νέο, σε νέο νομοθέτημα. Και αν χρειάζεται μια απλή πολιτική συνέχεια ή παρακολούθηση του θέματος. Ζητήσαμε τις απόψεις της, της ΟΚΕ, της Επιτροπής των Περιφερειών, του Ombudsman και μπορεί όλοι αυτοί να θέλουν να παρέμβουν. Δεν έχουν κάνει συγκεκριμένες επίσημες προτάσεις ώστε να εισαχθεί η ενδεχόμενη του συμμετοχή στη διαδικασία μέσα σε κάποιο σχέδιο, στο σχέδιο του κανονισμού, αλλά μπορεί και αυτό να μας απασχολήσει. Το ίδιο βέβαια και για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Διαπιστώσαμε στην ανταλλαγή με τα Εθνικά Κοινοβούλια πως τα ίδια δεν θέλανε να μπορούν να αναφέρονται στον κανονισμό. Αλλά Εν πάση περιπτώσει, για αυτό το δύσκολο και θεμελιώδη ζήτημα που πιθανότατα θα χρειαστεί να λυθεί αναπερίπτωση ανάλογα με τα θέματα και τις πρωτοβουλίε, αυτό το πρόβλημα δηλαδή της πολιτικής ε, παρακολούθησης, δηλαδή σε τι καταλήγουν τελικά όλα αυτά, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε πόσο σκοπεύουμε, τι είδου συνέχεια σκοπεύουμε να δώσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν σκοπεύουμε κάτι να κάνουμε πρέπει να το προβλέψουμε συγκεκριμένα στον κανονισμό ή αν αντιθέτω θεωρούμε πω η σιωπή του κανονισμού θα μα δώσει μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Λαμασούρ και εσείς μας κάνατε εξαιρετικά πλήρη και συγκεκριμένη και ξεκάθαρη παρουσίαση. Κατά λοιπά, να ευχαριστήσουμε και όλους τους εισηγητές. Όλους τους εισηγητές ε, γιατί μέχρι στιγμής έχετε δείξει μεγάλη ακρίβεια. Πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο. πρώτο και καλύτερο ο κύριο Εφνερ, που είναι και εισηγητή εξ ονόματο τη Επιτροπή Αναφορών. Παρακαλώ. liebe äh, Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ζήτα Γκουρμάη και ο Αλένα Μασούρ. παρουσίασαν την κοινή πρότασή τους τόσο διεξοδικά που δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Χρειαζόμαστε απλώ χρόνο για τη συζήτηση στην Επιτροπή. Είμαι ευγνώμων προς τους συνεισηγητές για την αγαστή αυτή συνεργασία. Είναι μια πρωτοφανής εμπειρία γιατί είναι η πρώτη φορά που τέσσερις συζητητές συνεργάζονται για την ίδια έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρόλο που από νομική άποψη έχουμε δύο εκθέσεις, μία έκθεση Επιτροπής Αναφοράς και μία έκθεση της αρμόδιας επί τη Επιτροπής που είναι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Πάντως η συνεργασία των τεσσάρων εισηγητών ήταν ε, ευθύ εξ αρχής στενή και θα συνεχιστεί προκειμένου να φτάσουμε σε κοινή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ε, διαβεβαιώ ότι μέχρι στιγμή η συνεργασία ήταν ε, θαυμάσια και ήταν πραγματικά απόλαυση αυτή η συνεργασία με τους συνεισηγητές. Ευελπιστώ ότι θα καταλήξουμε σε κοινέ θέσει με στόχο να διατρανώσουμε την ενωμένη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θα περιοριστώ στα σημεία που βρίσκονται στο επίκεντρο της δικής μας έκθεσης της Επιτροπής Αναφορών που συντάσσω από κοινού με την Ταϊάννα Γουόλης. Απλώς θέλω να κάνω και τις εισαγωγικές παρατηρήσεις για να εξάρω την αγαστή συνεργασία που είχαμε με τους δικούς σας συνεισηγητές. Είμαι πεπισμένος ότι θα καταλήξουμε σε κοινέ θέσεις για όλα τα σημεία και όλοι θα πλέψουμε προς την ίδια κατεύθυνση όπως συνέβη μέχρι τώρα. Το πιο σημαντικό σημείο για το οποίο υπάρχει μια μικρή διάσταση θέσεων είναι το θέμα των ακροάσεων και του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά τη γνώμη μας, είναι απαραίτητο να γίνουν αυτές οι δημόσιες ακροάσεις και να μην μπορεί να αποποιηθεί των ευθυνών της ή ε, να διαφύγει των ευθυνών της είναι να οργανώσει αυτές τις ακροάσεις. Άλλωστε δεν μιλούμε για ένα μηχανισμό άμεσης δημοκρατίας. Μιλούμε για έναν τρόπο λήψης αποφάσεων από τα κοινοτικά όργανα προκειμένου να λάβουν τις αποφάσεις ε, τους Μιλούμε για ένα μηχανισμό συμμετοχική και όχι άμεση δημοκρατία, όπου δίνουμε το δικαίωμα στου πολίτε να υποβάλουν προτάσει. Όπω είπε και ο Αλέλα Μασούρ, το δικαίωμα αυτό συνοδεύεται και από μια σειρά υποχρεώσεων. Υποχρεώσει που καλούνται να σεβαστούν οι Ευρωπαίοι πολίτε προ τον αριθμό των υπογραφών, τον αριθμό των χωρών τι οποίε συμμετέχουν, προθεσμίε κτλ. Πρόκειται για ένα μηχανισμό διαλόγου μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Και πιστεύουμε ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να αναλάβουν ε, και να πληρούν τις υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση που συλλεγούν ένα εκατομμύριο υπογραφές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να τηρήσει μια σειρά προϋποθέσεων. Οι παραλήπτες της πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων των πολιτών είναι υπεύθυνη και για την οργάνωση των δημοσίων ακροάσεων. Σε συνεργασία βέβαια και με τα άλλα θεσμικά όργανα, πιστεύουμε όμως ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλακεί ενεργά όπως και τα θεσμικά όργανα, αλλά σε καμία περίπτωση θα πρέπει να αποφύγει τις ευθύνες της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, διατύπωση της αιτιολογικής ε, σκέψης υπαριθμό 17 του σχεδίου που περιλαμβάνεται και στο διατακτικό στο άρθρο 11 παράγραφος Γ. Εκεί θεσπίζουμε διάφορες προθεσμίες. Πρώτη προθεσμία τριών μηνών για την εξέταση της πρωτοβουλίας πριν την διοργάνωση της ακρόασης και μετά μια προθεσμία δωδεκάμινη στη διάρκεια της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να λάβει μια απόφαση για το κατά πόσο θα δώσει συνέχεια, νομική συνέχεια στην πρόταση αυτών των πολιτών. Στη διάρκεια του δεκαμήνου αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε θα πρέπει να συμπεριλάβει τις προτάσεις στο πρόγραμμα εργασίας της για το επόμενο έτος ή να δικαιολογήσει για ποιο λόγο δεν κρίνει σκόπιμη τη συνέχεια αυτής της πρωτοβουλίας. Επαναλαμβάνω, υπάρχει μία μικρή διαφορά ως προς το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα, γιατί η Επιτροπή Αναφορών κρίνει ότι το 12 μήνο είναι πολύ στενό περιθώριο. Βέβαια, η διορία αυτή σχετίζεται και με την έννοια αυτή τη πρωτοβουλία. Γιατί δεν θέλουμε μια πρωτοβουλία για τα πολιτικά κόμματα. Και το λέω αυτό ανεπιφύλακτα. Αυτό ο μηχανισμό θα πρέπει να αξιοποιηθεί από του Ευρωπαίου πολίτε. Δεν θέλουμε ένα μηχανισμό που θα εξυπηρετήσει τα μεγάλα σωματεία ή του συνεταιρισμού στα κόμματα που ούτω ή άλλω είναι οργανωμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν δυνατότητα συγκέντρωση μεγάλου αριθμού υπογραφών. Εμεί θέλουμε ένα μέσο για νέε πρωτοβουλίε πρωτοβουλίες που πραγματικά θα εκπηγάζουν από τη βάση από τους Ευρωπαίους πολίτες και θα πρέπει να αξιοποιηθούν επικοδομητικά. Αν ήταν απλώς να δώσουμε ε, επιπλέον ευκαιρίες σε λόμπι και ομάδες πίεσης που ήδη εκπροσωπούνται στις Βρυξέλλες δεν θα ήταν μέσω συμμετοχικής ε, δημοκρατίας αυτό. Εμείς θέλουμε ε, ένα μέσο γιατί, και για αρνητικέ πρωτοβουλίε, για πρωτοβουλίε διαμαρτυρία εκ μέρου των πολιτών. Και είναι πολύ πιο εύκολο να συγκεντρωθούν υπογραφέ όταν ε, έχουμε μια πολιτική πρωτοβουλία. Πιο εύκολο δηλαδή είναι να συλλεγούν ταχύτερα υπογραφές για κάποια διαμαρτυρία. Τώρα, για την δυνατότητα να συμμετάσχουν οι πολίτες σε προτάσεις που θα πρέπει να έχουν και χαρακτήρα καινοτόμο, αυτό σημαίνει και μια δυνατότητα επικοινωνίας. Οι εμπειρίες που έχουμε μέχρι τώρα είναι οι πολύ σύντομες προθεσμίες, ότι, ότι οι πολύ σύντομες προθεσμίες στην ουσία παρεμποδίζουν. Και όταν μιλούμε και για το διεθνικό επίπεδο, εκεί η προθεσμία πρέπει να είναι ασφαλώς μεγαλύτερη από ότι μέσα σε μια ενιαία χώρα όπου συνήθως υπάρχει μια γλώσσα. Εδώ μιλούμε για με ένα πλήθο χωρών, με πολλέ διαφορετικέ γλώσσε και οι 12 μήνε σημαίνουν στην ουσία ότι όταν θα έχει παρέλθει το έτος αυτό και ίσω έχουν συλλεγεί 900.000 υπογραφέ, τότε αυτομάτω ακυρώνονται όλε αυτέ οι 900.000 υπογραφέ και δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα αφού δεν έχει φτάσει στο εκατομμύριο να επιτευχθεί ο απαιτούμενο αριθμό. Εμεί άλλωστε δεν βλέπουμε και κανένα αποχρόντα λόγο να πέφτει αυτή η δαμόκλειο σπάθη μετά από το έτος, από την πάροδο του έτους. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ του Κοινοβουλίου προτείνει στη γνωμοδότησή της 24 μήνες. Εμάς εν τέλει οι 18 μήνες μας φαίνονται α, λογικός συμβιβασμός. Αυτές οι διαφορές είναι όμως μάλλον λεπτές αποχρώσεις διαφορών μεταξύ ημών και εμείς βλέπουμε να ε, αποκρισταλώνονται ανάγλυφα τα επιχειρήματα εκατέρωθεν. Εμείς ήδη στην Επιτροπή Αναφορών το συζητήσαμε, στην ΠΕΤΗ, τώρα το συζητούμε εδώ στην Επιτροπή ΑΦΚΟ. Συνεργάζονται καλά οι εισηγητές και νομίζω ότι πρόκειται πραγματικά για ένα πείραμα που δείχνει ότι και στο μέλλον ε, σε σημαντικές επιτροπές θα μπορεί να γίνεται αυτή η διακομματική ε, συνεργασία. Θα αρκεστώ σε αυτά. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι παρουσιάστηκε το θέμα με εξαιρετικό τρόπο και χαίρομαι για οποιαδήποτε σχόλια έχετε και κριτική και διορθώσεις. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Νταφ, που είναι ο πρώτος στον κατάλογο αγοριτών, θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Σίγμουντ, που είναι η συγγήτρια της ε, Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και που ήδη ε, ήρθε στη συνεδρίασή μας τον Ιούλιο. Πάντως σας ευχαριστούμε που ξαναέρχεστε στην Επιτροπή μας, κυρία Σίγκμουντ. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με επιτρέπετε να συμμετάσχω. Ευχαριστώ και τους τέσσερις συζητητάς που μπόρεσα να συζητήσω μαζί τους. Χαίρομαι που το αίτημά μας στην ουσία και οι στόχοι μας ταυτίζονται. Συμφωνώ απολύτως με την άποψη που ακούστηκε ότι δεν πρόκειται για μηχανισμό άμεσης δημοκρατίας αλλά περισσότερο για μια δυνατότητα να κινητοποιηθούν οι πολίτες. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μηχανισμών κατά χάμπερ μας, δηλαδή δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, πρόκληση κοινών συζητήσεων και θετικό επηρεασμό των πολιτών. η Επιτροπή μας λοιπόν, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να συμβάλλει, να παρακινήσουμε λοιπόν νέα στρώματα δραστηριών πολιτών να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πρόταση της Επιτροπής σας ΑΦΚΟ στον τομέα της ε, δραστηριοποίησης των θεσμικών οργάνων νομίζω θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και η Επιτροπή μας θα βοηθήσει να ε, λάβουμε απόφαση για το πώς θα συμμετάσχουμε. Εσείς κύριε Ντάφ. Ευχαριστώ όλους όσοι εξήγησαν τις απόψεις τους. Έχω ερωτήσεις και σχόλια ωστόσο. Πρώτο. Τροπολογία 4. αριθμός κρατών από τα οποία θα πρέπει να συλλεχθούν οι υπογραφές. Η συνθήκη λέει ότι θα πρέπει να προέρχεται από σημαντικό αριθμό κρατών. Μόνο αυτό λέει. Και είχαμε πει και κατά την σύνταξη της συνθήκης ότι θα το βάλουμε αυτό επίτηδες διότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε πολυεθνικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας αυτής. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι το 1 πέμπτο των χωρών μελών είναι σημαντικός αριθμός. Θα προτιμούσα να εμείνουμε στο 1 τρίτο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξάλλου, θεωρώ ότι είναι παράδοξο ότι οι συγκητές φαίνεται να προτείνουν ένα πέμπτο των χωρών από τις οποίες να προέλθουν υπογραφές αλλά σε ό,τι αφορά την οργάνωση της Επιτροπής Πολιτών ξαφνικά μιλούν για επτά χώρες. Το πέμπτον του 27 είναι 6 ωστόσο. Δεν βλέπω λοιπόν πώς γεφυρώνεται αυτή η διαφορά. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Πολιτών, τροπολογία 6, δυστυχώς εξακολουθώ να μην κατανοώ γιατί άρα γι' αυτό να είναι απαραίτητο. Η συνθήκη τηρεί σιγή σε ό,τι αφορά την οργάνωση. Μιλεί μόνο για ένα εκατομμύριο πολιτών. Μου φαίνεται ότι η επιβολή Επιτροπής Πολιτών Επτά πολιτών από επτά χώρες, χώρες μέλη, μου φαίνεται λοιπόν απολύτως περιττή. Απολύτως περιττό φίλτρο ή κατόφλι, αν θέλετε, που εξάλλου θα απαιτήσει παράγω δίκαιο θέσπιση παραγωγού δικαίου για να νομιμοποιείται αυτή η Επιτροπή, θα σημάνει περαιτέρω καθυστερήσεις της διαδικασίας, καθώς και περαιτέρω γραφειοκρατικά κολλήματα. Πολιτικοποιημένα ή κομματικοποιημένα συνδικάτα ή επαγγελματικές οργανώσεις δεν θα διστάσουν να αρπάξουν την ευκαιρία αυτή ή να πω αλλιώς να ξεπεράσουν εύκολα το κόλλημα αυτό, αλλά ο απλός πολίτης θα βρει εξαιρετικά μεγάλες δυσχέρειες για να βρει άλλους έξι απολύτως άγνωστούς του από έξι χώρες μέλη για να συνδυάσει προσπαθίες του μαζί τους. Δεν νομίζω ότι οι σωστές πρωτοβουλίες ξεκινούν από μια επιτροπή. Ε, εκτός βέβαια από την Συνταγματική Επιτροπή. Τροπολογία 12 λέει εν απουσία, λήψη μάλλον αρμοδίας εκλογικής αρχής της Ένωσης. Η πρότασή μου είναι να δημιουργηθεί τέτοια εκλογική αρχή. και να συνδυαστεί και μια πρόταση για την θέσπιση της αντίστροφης αναλογικότητας για την θέσπιση της. Είναι λοιπόν δύο σημαντικά νομοθετήματα που πρέπει να κινηθούν παράλληλα. ερωτήσεις. Τι θα γίνει εάν μια πρωτοβουλία προτείνει ανάληψη νομικής πρωτοβουλίας της Ευρωβουλής. Σε το μισό που το Κοινοβούλιο χέρι του προνομίου πρωτοβουλίας. Η ίδια αμφισημία θα υπάρξει και στην περίπτωση του Συμβουλίου όπου ορισμένες χώρες μέλη μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλία με την κατάθεση σχεδίου νόμου για θέματα εσωτερικής, εσωτερικών υποθέσεων και δικαιοσύνης. Θα αποκλείσουμε τους ευαίσθητους αυτούς τομείς που ενδιαφέρουν τους πολίτες. και όπου Συμβούλιο και Κοινοβούλιο έχουν ίδιο δικαίωμα πρωτοβουλίας. Ο Δε Λαμασούρ είπε ότι έκκληση για τροποποίηση της συνθήκης δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πρωτοβουλίας πολιτών ερμηνεύοντας αυστηρά τη συνθήκη, αυτό είναι σωστό, αλλά θα είναι δύσκολο να το εξηγήσει κανείς στους πολίτε που γνωρίζουν ότι η Κομισιόν αλλά και ιδίω το Κοινοβούλιο έχουν το δικαίωμα να προτείνουν αλλαγή στη συνθήκη. Θα είναι πρόβλημα να εξηγηθεί στους πολίτες, κανένα εκατομμύριο πολίτες, ότι η πρωτοβουλία τους είναι άκυρη και ανυπόστατη, ενώ αυτό που ζητούν είναι κάποια εύλογη αλλαγή στην συνθήκη. Εν τέλει, τι γίνεται εάν μια πρωτοβουλία απαιτεί αλλαγή του δημοσιονομικού σχεδιασμού της Ένωσης, αλλαγή των δαπανών που να ξεφεύγει από τα όρια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Τι πράττει τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν καταχωρίζει τέτοια πρωτοβουλία. Ενώ θα μπορούσε να έχει ένα απολύτως εύλογο χαρακτήρα μια τέτοια πρωτοβουλία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με τη σειρά μου θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους τους συζητητές και να τονίσω ότι έχει γίνει σοβαρή και εντατική δουλειά με ακροάσεις σε όλες τις πολιτικές ομάδες, με διάφορες διαβουλεύσεις, όπως είπε και η κυρία Γκουρμάη, με οργανώσεις και ούτω καθεξής και εκτός Ευρωβουλής. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό το Κοινοβούλιο ασχολείται εντατικά και με τρόπο θα έλεγα επιθετικό με την πρωτοβουλία αυτή και δημιουργεί έτσι μια διασύνδεση με την δημόσια συζήτηση που γίνεται. Όπως είπε η κυρία Κουρμάη, με την ατυχή αυτή δυστυχώς μεγάλη αποχή στις ευρωεκλογές οφείλει κανείς να σκεφτεί με ποιον τρόπο μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το έλλειμμα δημοκρατικότητας στην ε, ευρωπαϊκή πολιτική ζωή και πώς μπορούν να παρακινηθούν οι πολίτες να συμμετάσχουν περισσότερο. Στην πρόταση ψηφίσματο και σε ό,τι αφορά τι τεχνικές προδιαγραφέ και τι συνθήκε και όρου. και εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να διατεθούν όσο, γίνεται, όσο γίνεται περισσότερες δυνατότητες υπέρ των πολιτών, χαμηλά κατόφλια, ώστε να νιώσουν οι πολίτες ότι αναμειγνύονται στην πολιτική. Ένα θέμα που για μένα είναι σημαντικό και όπου θίγεται η ουσία και αναφέρομαι στην τροπολογία υπαριθμών 7 και που στην μέχρι τώρα συζήτηση έχει παίξει σημαντικό ρόλο, δηλαδή οι σχέσεις μεταξύ άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε λίγο, διότι βέβαια οι προσδοκίες των πολιτών από την ευρωπαϊκή πολιτική έχει πάντοτε σχέση με την προσωπική ευημερία, με την προσωπική αντίληψη του τι σημαίνει δημοκρατία για τον καθένα. Δεν βρισκόμαστε σε κάποιο χώρο εκκρεμής, αλλά υπάρχουν άμεσες επιπτώσεις στην εθνική πολιτική ζωή και οι πολίτες κάθε χώρας θίγονται από τις πολιτικές αποφάσεις και εντάσσονται μέσα σε ένα δίκτυο διασυνδέσεων και επιτέλους σκέπτονται έχω την δυνατότητα να επηρεάσω το πολιτικό γίγνεσθε. Το πολιτικό γίγνεσθε. Και νομίζω οι προσδοκίες από το μηχανισμό που συζητούμε είναι τόσο μεγάλες που εάν δεν καταστήσουμε σαφές ότι δεν πρόκειται για μηχανισμό άμεσης δημοκρατίας αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ανοίξουμε δυνατότητες όπου οι πολίτες αμφωτέρων των φύλων να μπορούν να εκφράσουν τη δυσαρεσκιά τους με την πολιτική όπως αυτή ασκείται στο ευρωπαϊκό επίπεδο, να διασυνδέσουν αυτήν την έκφραση με πρωτοβουλίες, που σημαίνει ότι πρέπει ίσως στο ίδιο το ψήφισμα να περιλάβουμε μία παράγραφο που να φύγουμε ακριβώς αυτό το θέμα αυτής της φαιάς ζώνης που διαγράφεται να πούμε δηλαδή ότι υπάρχουν θέματα τα οποία δεν καλύπτονται από τους μηχανισμούς της ε, συνθήκης Λισαβόνας που έχουν όμως απολύτως θεμητό χαρακτήρα όπως, τον, όπως αισθάνονται τις συνέπειες, δηλαδή τις επιπτώσεις της πολιτικής οι ε, πολίτες. Και υπάρχουν πράγματι ε, εκπρόσωποι και στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή που σκέπτονται ότι ίσως μπορεί η σημερινή οικονομική κρίση να ξεπεραστεί και με μια τροποποίηση τη συνθήκης ή μια τέτοια να συμβάλλει σε αυτήν. Και μιλώ για θέματα όπως δημοσιονομική εποπτεία κλπ. Εξού και προτείνω, όπως είπα, να περιλάβουμε ένα εδάφιο που να καταστά σαφές ότι θέματα τα οποία δεν καλύπτονται από τους υφιστάμενους μηχανισμούς θα είναι δυνατόν να προβάλλονται και τότε πλέον Συμβούλιο και Κοινοβούλιο είναι αυτά που λαμβάνουν την εντολή να καταστήσουν ίδιες τις θέσεις αυτές και με τη σειρά τους με συμμετοχή ή με λήψη υπόψη των θέσεων αυτών των πολιτών να αναλάβουν πλέον αυτά τα ίδια τα θεσμικά όργανα πρωτοβουλίες και να απευθυνθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε νομίζω οξύνεται περισσότερο ο μηχανισμός αυτός και καλύπτει έτσι θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν καλύπτονται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Διαφαίνεται ανάγκη διοργάνωση των εργασιών μας, διότι πρέπει να κλείσουμε τις εργασίες στις 12.30. Εγώ έχω έξι ακόμα μιλητές εδώ. Μετά πρέπει να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Επιτροπής και να μπορέσουν να απαντήσουν και οι εισηγητές, Λαμασούρ και Γκουρμάη. Κατά συνέπεια, πρέπει να κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών, να διαβάσω ποιοι είναι. Κλείνω λοιπόν τον κατάλογο των ομιλητών. Εντάξει. Θα πρέπει να σας πω ότι με έναν απλό μαθηματικό υπολογισμό δεν μπορώ να δώσω παρά τρία λεπτά στον καθέναν. Λοιπόν, τρία λεπτά η συνάδελφος για τεμάκι. Sorry, I didn't hear. Thanks. Uh, I try to be very... Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Χαίρομαι για την αγαστή συνεργασία μεταξύ των συνεισηγητών, γιατί όπως είπε ο κ. Λαμασούρ, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συγκεντρώσουμε την ε, ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία υπέρ της έκθεσης. Έχω μερικά σχόλια για την διαπραγματευτική εντολή, όπως λέει το έγγραφο. Νομίζω ότι ο στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει είναι να είναι όσο πιο εύχρηστη και πιο απλή γίνεται η πρωτοβουλία αυτή των πολιτών και όσο πιο φιλική γίνεται προς τους πολίτες, προς τους χρήστες. Οπότε, γι' αυτό και ο έλεγχος του παραδεκτού θα πρέπει να γίνεται σε όσο το δυνατό ε, πρόωρη φάση γίνεται. Όσο πιο νωρίς γίνεται, γιατί αν γίνει αυτός ο έλεγχος σε προχωρημένο στάδιο, η κατάσταση που θα δημιουργηθεί θα είναι δυσάρεστη. Αναφέρεται στο σημείο 4 ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει όσο το δυνατόν λιγότερες προσωπικές πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται ούτε αριθμός διαβατήριου, ούτε αριθμός ταυτότητας στην καταγραφή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό οι αποφάσεις περί παραδεκτού να υπόκεινται σε ένδικο μέσο μόνο ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβήτη. Αν υπάρχουν φυσικά ε, βάσιμοι λόγοι για κακή διοίκηση. Αυτό είναι σημαντικό και για την Επιτροπή και για το Κοινοβούλιο. Έχω και δύο προσωπικά σχόλια. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Νταφ ότι η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να αφορά και πρόταση για αλλαγές στη συνθήκη. Και μάλιστα συντάξω και σχετική τροπολογία για το θέμα αυτό. Η δεύτερη προσωπική μου γνώμη είναι ότι είναι Κρίμα να περιορίζουμε τις υπογραφές μόνο στους πολίτες και όχι στους κατοίκους. Είναι θέμα ισότητας, αλλά και πρακτικό ζήτημα. Γιατί αν συγκεντρώνουμε τις υπογραφές και έχουμε και κάποιους κατοίκους που θέλουν να υπογράψουν, αλλά δεν μπορούν. γιατί μόνο οι πολίτες δικαιούνται να υπογράψουν. Οι υπήκοοι δηλαδή. Γιατί να το περιορίζουμε μόνο στους υπηκόους. Θα ήθελα να το ξανασυζητήσουμε αυτό. Σας ευχαριστώ, κυρία Κοράτσα. Μπορείτε να μιλήσετε ποια γλώσσα θέλετε, αφού είστε πολύ γλώσσα. αλλά φιλανδικά όχι. Όμως θέλετε Μιλήστε τη δική μου γλώσσα, θα είμαι πολύ περήφανος. Διαφορετικά, όποια άλλη θέλετε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ευχαριστεί που ακόμα και ένας Ιταλός λέει διαφορετικά το όνομά μου. Ε, εγώ θα μιλήσω στα αγγλικά και θέλω να σας συγχαρώ τους εισηγητές και εσάς Πρόεδρε που δείχνετε τέτοιο ανοιχτό πνεύμα και συμμετοχή ήδη στη διαδικασία. Εγώ ως εισηγήτρια στην ΛΥΜΠΕ για το ΕΛΚΑ είχα την ευκαιρία να εκφράσω τις απόψεις μας ε, και εκτιμώ ιδιαίτερα τη σημερινή αυτή συνάντηση. Στη ΛΥΜΠΕ συζητήσαμε δύο πράγματα, υπέρ μάλλον δύο πραγμάτων που, που θα ήθελα να σας ζητήσω να στηρίξετε κι εσείς. Αρχίσω από το πιο απλό. Στο πνεύμα αυτού του το ανοιχτό για συμμετοχή και για προσβασιμότητα στους πολίτες, να σκεφτούμε όχι μόνο το κριτήριο της μόνιμης διαμονής, αλλά και της εθνικότητας. Έτσι ώστε να μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν σε τρίτες χώρες να έχουν πρόσβαση στο μέσο αυτό. Κατά την άποψή μας είναι το άρθρο 7, είναι μια τροπολογία που πέρασε στην Λίμπε και λέει ότι ότι το πρώτο κριτήριο θα πρέπει να είναι η διαμονή, αλλά θα πρέπει να μπορεί να εξεταστεί και επί τη βάση της εθνικότητας. Και αυτό για να λύσουμε κι άλλο ένα πρόβλημα. Α πούμε για το Βέλγιο. Υπάρχουν τεράστιοι ε, αριθμοί μη Βέλγων πολιτών που ζουν στι Βρυξέλλε, για παράδειγμα. Εκείνοι άμεσα θα κάλυπταν την ποσόστοση των Βέλγων αν, ληφθούν υπόψη μόνο, αν ληφθεί υπόψη μόνιμη διαμονή τους. μένει από εμά είμαστε τέτοιου είδους πολίτε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σκεφτείτε πρώτον την διαμονή τη μόνιμη διαμονή και δεύτερον την εθνικότητα. Το δεύτερο ζήτημα είναι πιο περίπλοκο και είναι το θέμα της διαφάνειας. Είμαστε υπέρ των όσων είπε ο κύριος Λαμασούρ και των όσων και εσείς συμφωνείτε ότι θα πρέπει να ισχύουν, ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μέγιστη οικονομική διαφάνεια. Εγώ θα ήθελα να στηρίξω ότι θα έπρεπε να απαγορεύεται να δίνεται χρηματοδότηση από τις πολιτικές ομάδες και πολιτικά κόμματα. Θα χρησιμοποιήσουμε το ΑΕΛΚ ή άλλες, ε, ε, ε, τα χρήματα άλλων ομάδων για να χρηματοδοτήσουμε τέτοιου είδους εκστρατείες για τις πρωτοβουλίες των πολιτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τεθούν κάποια όρια, γιατί έτσι θα μπορούμε να δώσουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα στους πολίτες ότι είμαστε πολύ σταθεροί κατά οποιασδήποτε πιθανή μορφή κατάχρησης για δικούς μας πολιτικούς στόχους. Και θα ήθελα να σας καλέσω να στηρίξετε την ε, τροπολογία που ψηφίστηκε στη Λίμπε ω προς αυτό. Τρίτο σημείο που κατά την άποψή μου είναι το πιο σημαντικό έχει να κάνει με τη σχέση ανάμεσα στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία και ανάμεσα στη δημοκρατία. Η... Βεβαίως, σε σχέση... το, το γεγονός ότι δεν πρόκειται για νομοθετική πρωτοβουλία και αυτό παραμένει στα χέρια της Κομισιόν και πρόκειται για πολιτική ε, πρωτοβουλία. Αν όμως 7-8 από εμά μπορούμε να οργανωθούμε και να κάνουμε μια πρωτοβουλία, Πού είναι οι πολίτε, ποιο είναι το νόημα. Εμεί και εμεί είμαστε πολίτε, ναι, εντάξει, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να εκφραστούμε μέσω τη ε, Δημοκρατία, τη δημοκρατική εκπροσώπηση. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί όμω και θέλουμε να στείλουμε ένα σοβαρό πολιτικό μήνυμα στου πολίτε και ότι ναι όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε εδώ και έξι μήνες που μιλάμε και λέμε ότι θέλουμε να είναι πιο, προς, πιο, ε, πιο προσιτή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τότε δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε εκλεγμένου πολιτικού να οργανώνουν μια πρωτοβουλία των πολιτών. Εντάξει, μπορούν να το υπογράψουν και να το στηρίξουν ή εν πάση περιπτώσει να το συζητήσουν, αλλά να μην ξεκινάνε οι πρωτοβουλίε από εμά. Γιατί κάτι τέτοιο θα, θα, θα εκφυλίσει τον στόχο που θέλουμε να πετύχουμε. Ολοκληρώνετε παρακαλώ γιατί έχετε περάσει τα τρία λεπτά. Ναι, ναι, ολοκληρώνω. Υπάρχει λοιπόν τέτοια τροπολογία που πέρασε στη Λίμπε και σας καλώ να την στηρίξετε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος Μπρόνς. Ευχαριστώ. Ο όρο πρωτοβουλία των πολιτών προποθέτει ε, ότι η εξουσία για το περιεχόμενο οποιασδήποτε πρόταση επαφίεται στου πολίτε. Όταν οι πολίτε ψηφίζουν σε ένα δημοψήφισμα ή στι εκλογέ, ανταποκρίνονται σε μία περιορισμένη ερώτηση. Μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ενό ναι ή ένα όχι, ενώ μεταξύ ενός υποψηφίου ή ενός άλλου, αλλά η πρωτοβουλία των πολιτών είναι ενό διαφορετικό. Η ενό αλλου αλλα η πρωτοβουλια των πολιτων ειναι κατι διαφορετικο η διατυπωση και ο τρόπος δράσης κανονικά επαφείται στου πολίτες, στους κυβερνόμενου και όχι στους κυβερνώντε. Βέβαια αυτό δεν είναι ε, απόπειρα να δοθεί σε ανώνυμους πολίτες το δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας, αλλά να τους επιτρέψει να πούν αυτό που τους επιτρέπεται να πούν και να κάνουν. Στο άρθρο 4 της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ότι οι πρωτοβουλίες που δεν είναι σοβαρές, θερούνται σοβαρότητες, δεν ξέρω ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, ή ε, στην παράγραφο 4 είναι κατάφορα παραβιάζουν κατάφορα αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύονται. Αυτό όμω είναι υποκειμενικά. Έχουμε την αξιοπρέπεια, σοβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά είναι καλά. Οι περισσότεροι αποκαλούνται δημοκράτες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρόλο που συχνά περισσότερο ενδιαφέρονται για τα δικά τους δημοκρατικά δικαιώματα και των φίλων τους και όχι των αντιπάλων τους. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για ανθρώπινα δικαιώματα, εννοεί τον άλλον των ομοειδεατών, όχι των αντιπάλων της, των ιδεολογικών. Το δικαίωμα πρώτες πρωτοβουλίες των πολιτών είναι ουσιαστικά δικαίωμα μόνο να συμφωνήσει κανείς με το ευρωπαϊκό σχέδιο. Μπορεί να προτείνει ο πολίτης, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αρνηθεί να δώσει συνέχεια. Οπότε ουσιαστικά δεν δίνουμε περισσότερη εξουσία στους πολίτες από ό,τι δίνουν οι εφημερίδες στους πολίτες που μπορούν να στείλουν επιστολές σε μια εφημερίδα αλλά ο συντάκτης αποφασίζει αν θα τη δημοσιεύσει ή όχι. Δεν είναι συμφωνία συνεργασίας ε, παρά μόνο ε, συμφωνία να χειροκροτήσει, να συμφωνήσει και να επικροτήσει. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαφωνίας. Εγώ είμαι υπέρ του περιορισμού του αριθμού των χωρών και την πρόληψη των υπογραφών. Είμαι υπέρ της ηλεκτρονικής συγκέντρωσης υπογραφών και της, του περιορισμού του χρονικού περιθωρίου. Παρ' όλα αυτά, οι πρωτοβουλίες μπορεί κάλλιστα να πνιγούν στα σπάργανα και υποκειμενικά, αν είναι αντίθετες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μια και έχουμε περιορισμένο χρόνο αγόρευση, θα επικεντρωθώ στα ουσιώδη σημεία. Καταρχήν, η Επιτροπή των Πολιτών. Σημείο 1. Δεν αναφέρεται ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο εκθέσεων της Επιτροπής ΑΦΚΟ και τη Επιτροπή Αναφορών. Λέμε ότι στη μία έκθεση 7 ή 8 εκπρόσωποι διαφορετικών χωρών θα πρέπει να συμμετέχουν, ενώ στην Επιτροπή Αναφορών αναφέρονται 7 εκπρόσωποι από τρει χωρε Στη, η μία επιτροπή ζητά 7 χωρε και η άλλη αρκείται σε 3. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ υπερβολική η απέτηση τη Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Οι 7, εκπρόσωποι, 7 μέλη τη επιτροπή να εκπροσωπούν να προέρχονται από 7 διαφορετικέ χώρε. Επίση, για το θέμα τη καταγραφή η πρόταση της Επιτροπής Σταγματικών Υποθέσεων είναι πιο ήπια από την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πιο αυστηρή. Εγώ είμαι μέλος της Νομικής Επιτροπής και μας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα των νομικών βάσεων, γι' αυτό θα ήθελα να σας κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου. Θα πρέπει να επισημάνουμε μία νομική βάση. Γιατί είναι πολιτικός ο χαρακτήρας ε, αυτής της πρωτοβουλίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με την Κύπρο, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τελείως το θέμα της νομικής βάσης. Επίσης, το θέμα της εξακρίβωσης των υπογραφών. Εγώ είμαι υπέρ τη πρώτη Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και όχι τη Επιτροπή Αναφορών. Να αναφέρεται απλώ δηλαδή το όνομα και ο τόπο κατοικία και η υπογραφή. Εγώ ω συμβολογράφο Διαφωνώ γιατί στη Γερμανία ειδικά, στο Νότο, στη Βαβαρία, έχουμε περιπτώσεις όπου ο γιος έχει το ίδιο ονοματεπώνυμο με τον πατέρα και μέχρι τα 19 μπορεί να συγκατοικεί με τους γονείς του, να μένει ακόμη στο πατρικό και είναι πολύ δύσκολο να εξακριβώνουμε τις υπογραφές. Πρέπει να ακούμε σε δείγματα, δεν μπορούμε να εξακριβώνουμε όλες τις υπογραφές. Για παράδειγμα, είχαμε μια περίπτωση όπου ο γιος που έφερε ίδιο ονοματεπώνυμο με τον πατέρα είχε πωλήσει αγροτεμάχια του πατρό του. Επίση αν ανοίξετε ένα τηλεφωνικό κατάλογο, βρίσκεται εκατοντάδε Χαν Σμιτ. Σίγουρα θα υπάρξουν ε, διπλές υπογραφές αν χρησιμοποιήσουμε μόνο τη δειγματοληψία. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται και ημερομηνία γέννηση, για να μην πω και τόπος γέννησης. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό ταυτότητας, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη και αυτή την κατάσταση, αλλά στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει ταυτότητα, δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητα, θα πρέπει να αρκεστούμε στον αριθμό της ε, κοινωνικής ασφάλισης. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν τι χρειάζονται για τον προσδιορισμό της ε, ταυτότητας αν αρκεστούν στην, στον αριθμό της ταυτότητας ή στον αριθμό της κοινωνικής ασφάλειας για παράδειγμα, από ορισμένε. χώρες. Συμμετείχαμε σε πολλά δημοψηφίσματα στο Βερολίνο και πολύ συχνά έχουμε ένα εξάμεινο για τη σύλλογη των υπογραφών. Αυτό όμως ε, δημιουργεί και ένα πρόβλημα στη νομική βάση, γιατί έξι μήνες ε, είναι αρκετό διάστημα, αλλά δωδεκάμινο είναι υπερβολικό χρόνος. Τι θα γίνει αν μετά από 15 μήνε κάποιο ανακαλέσει την υπογραφή του επειδή η κατάσταση έχει αλλάξει η νομική ή άλλη. Και ίσως έχουμε το πρόβλημα παράλληλης κίνησης πλειώνων πρωτοβουλειών πολιτών, 5 και 6, που θα υπάρχει επικάλυψη χρονικά. Αυτό που θα πρέπει να γίνεται είναι να διεκπεραιώνονται αυτές οι πρωτοβουλίες πολιτών ή δυνατόν η μία μετά την άλλη. Άρα εγώ θεωρώ ότι η προθεσμία δεν πρέπει να υπερβαίνει του 12 μήνες. Σωστό είναι επίση αυτό που λέει η Επιτροπή Πετή, αναφορών δηλαδή, να γίνεται ακρόαση των ενδιαφερομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το πέρα συλλογή των υπογραφών. ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ ειλικρινά όλους τους εισηγητές των επιτροπών που συμμετείχαν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω ιδιαίτερος τον κύριο Λαμασούρ και την κυρία Γκουρμάη, γιατί ήταν πραγματικά και οι δύο η ψυχή αυτής της έκθεσης της Επιτροπής Σταγματικών Υποθέσεων. Το συνταγματικό δίκαιο και οι πολιτικές επιστήμες προβλέπουν ότι όταν θεσπίσετε ένα δίκαιο θα πρέπει να περιορίζετε κιόλα. Και θα ήθελα να σας συγχαρώ στην περίπτωση αυτή, γιατί καταφέρατε να ρυθμίσετε αυτό το δίκαιο με, τις λιγότερες δυνατές, με τους λιγότερους δυνατούς περιορισμούς. Και αυτό ανταποκρίνεται στην, στη φιλοδοξία μας να ενισχύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες και να τους αναδείξουμε ως πρωταγωνιστές της διαδικασίας της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Θα ήθελα να σας επισημάνω δύο σημεία για τα οποία καλό θα ήταν να εμβαθύνουμε τη σκέψη μας. Ένα από αυτά είναι η προσπάθεια αποφυγής ή στο θέμα του παραδεκτού μη αποδοχής πρωτοβουλειών που αντιβαίνουν σε προηγούμενη διάταξη και του κοινοτικού δικαίου. Δηλαδή, για να αποφύγουμε αυτή τη σύγκρουση νομιμοποίησης μεταξύ της συμμετοχικής δημοκρατίας και της ε, αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας θα πρέπει να προσδιορίσουμε ότι όταν δρομολογείται μία πρωτοβουλία της Επιτροπής ή του Συμβουλίου ή όταν πρόσφατα έχει θεσπιστεί κανονισμός ή νομοθετική διάταξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει για ένα μικρό διάστημα να περιορίσουμε αυτή την πρωτοβουλία για να μην εκλειφθεί ως προσπάθεια αντίθεσης ή κατάρριψης προηγούμενης νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι απόλυτη αυτή η διάταξη, είναι προσωρινή. Θα μπορούσε κάλλιστα να υποβληθεί μια τέτοια πρωτοβουλία, αλλά αργότερα, όχι αμέσως μετά την έγκριση με συγκεκριμένη διάταξη. Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά κόμματα και την Οργανωτική Επιτροπή, νομίζω ότι έχει νόημα η Οργανωτική Επιτροπή να μην απαρτίζεται από οργανικές δομές πολιτικών κομμάτων ή από άμεσα ή έμεσα όργανα των πολιτικών κομμάτων. Βέβαια, δεν μπορούμε να στερήσουμε από κάποιον τη δυνατότητα να συμμετέχει σε μια οργανωτική επιτροπή μόνο και μόνο επειδή είναι μέλος ενός συγκεκριμένου κόμματος. Αυτό θα ήταν πραγματικά η παραβίαση του δικαιώματος ε, ε, του συνεταιρίζεσαι ή τη συμμετοχή σε συγκεκριμένο κόμμα όχι όμως τα πολιτικά κόμματα να συμμετέχουν ε, ως τέτοια σε οργανωτική επιτροπή, ούτε αρχηγοί κομμάτων, αλλά μέλη κομμάτων κάλλιστα θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε μια οργανωτική επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ταρκόφσκι. Καταρχήν συγχαρητήρια στους εισηγητές για την πολύ καλή δουλειά τους. Πιστεύω πως τα αποτελέσματα της δουλειά αυτής, όπως είπε ο Λέν Λαμασούρ στην εισήγησή του, είναι να ε, γίνει αυτή η δυνατότητα πιο φιλική προς τους πολίτες. Εγώ δεν θα ήμουν τόσο αυστηρό ε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο κάποιοι συνάδελφοι ε, που είπαν ότι η αρχική πρόταση ήταν εκεί για να αποκλείσει, να μπλοκάρει αυτή την πρωτοβουλία Σίγουρα μπορεί η Κομισιόν να επιβαρυνθεί πολύ, αλλά νομίζω πως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι και όντως να καταστήσουμε αυτή τη δυνατότητα πιο ωφελική προς τους πολίτες. Και ένα από τα σπουδαία παραδείγματα για το πώς τα κατάφεραν οι εισηγητές μας είναι όταν πρόκειται για την καταγραφή και την πληροφορίες για μια τέτοια πρωτοβουλία. Γιατί η, προβο... η Κομισιόν πρότεινε την νομική βάση. Ξέρουμε πως ακόμα και οι νομικοί τσακώνονται μέσα στα θεσμικά όργανα για την νομική βάση. Ακούστηκαν και στην Νομική Επιτροπή κάποιες φωνές που για διαγραφή αυτή τη προπόθεση, αλλά τελικά συμφωνήσαμε για την ε, κατάλληλη διάταξη της συνθήκης. Και νομίζω πως αυτή είναι μια πολύ καλή συμβιβαστική λύση γιατί υποδεικνύει την προσέγγιση μας ε, έτσι ώστε να μην είναι τόσο δύσκολο όσο κάποιες φορές είναι στις προτάσεις της Κομισιόν, αλλά να είναι με φιλικό για τους, τους πολίτες, αλλά από την άλλη πλευρά να υπάρχει και κάποια ευθύνη που θα βαραίνει τους ίδιους τους πολίτες, γιατί είναι πολύ σημαντικό και οι πολίτες όταν θα κάνουν προτάσεις να συνειδητοποιούν αν μπορεί αυτό να είναι σχετικό με τις συνθήκες ή όχι. Γιατί όλοι θέλουμε να γίνει αυτό, αλλά κατά κάποιο τρόπο να μας επιτρέψει να μπούμε και σε μια συζήτηση για το ποιες είναι οι συνθήκες της συνθήκης, τι μας επιτρέπει ακριβώς να κάνουμε η συνθήκη. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα όσον αφορά αυτό το διάλογο μεταξύ θεσμών και πολιτών. Για την τροπολογία 39 θέλω να κάνω ένα σχόλιο που λέει ότι οι υπογράφοντες που έχουν μόνιμη κατοικία σε μια τρίτη χώρα θα θεωρηθεί πω προέρχονται από τις χώρες μέλη των οποίων είναι υπηκόοι. Έχω κάποιε ερωτήσει εδώ και ορισμένοι το ερμήνευσαν και λάθο ότι μπορεί να πρόκειται για ανθρώπου που δεν είναι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω πως θα πρέπει να δουλέψουμε για αυτή τη διάταξη ώστε να είναι σαφέστερη. Και όταν λέμε πολίτες Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν ε, μόνιμη κατοικία, μόνιμη διαμονή σε μια τέτοια χώρα θα πρέπει να είναι ε, πιο ξεκάθαρο και να μην λέμε μόνο οι υπογράφοντε, γιατί αυτό μπορεί να είναι παραπλανητικό. Ευχαριστώ, ήταν απλά ένα σχόλιο. Σας ευχαριστώ. Ε, κλείσαμε τον κατάλογο των ομιλητών, αλλά θέλετε να παρέμβετε. Αν είστε σύντομος, ναι. Όχι, απλώς θέλω να πω ότι οι συνεισηγητές μας είχα ζητήσει μια άτυπη εντολή για να συζητήσουμε μεταξύ τους εν ώψη της ε, ψηφοφορίας που θα γίνει στην Επιτροπή. Μετά τη σημερινή συζήτηση όμως και μετά το πνεύμα που επικράτησε, νομίζω ότι μπορούμε κάλλιστα να τους ε, χορηγήσουμε αυτή την άτυπη εντολή, αρκεί να μας ενημερώνουν τακτικά για την πορεία. Βεβαίως, ε, για αυτό το θέμα. Το είχα μάλιστα πει στην αρχή το θεωρούσα δεδομένο. Νομίζω και ο συνάδελφος Νταφ όμως αρνητικά είναι διακείμενος. Ναι, φοβούμαι ότι δεν πιστεύω πως η Επιτροπή μας θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Με όλο το σεβασμό, η συζήτηση σήμερα άνοιξε διάφορα σημαντικά μέτωπα που πρέπει να συζητηθούν εδώ στην Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι, για παράδειγμα, η δεύτερη παράγραφος του σχεδίου εντολής που μιλά για την Επιτροπή Πολιτών ή επτά ανθρώπους από επτά διαφορετικά κράτη ε, βρίσκει σύμφωνη την πλειοψηφία της Επιτροπής. Νομίζω επίσης ότι υπάρχει διαφωνία και για την παράγραφο 3 που αφορά το κατόφλι του αριθμού των κρατών μελών. Και ειλικρινά, με όλο το σεβασμό στους δύο συνεισηγητές, υποψιάζομαι πως δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Και ούτε καν θα πρέπει να προσπαθήσουμε. να βιαστούμε, να πάμε δηλαδή στο fast track στην πρώτη ανάγνωση. Νομίζω πως χρειάζεται χρόνος και χώρος για να υποβάλουμε τροπολογίες. Και να εξετάσουμε και πάλι σοβαρά το θέμα. Εντάξει, ωραία και καλά ότι συμβουλεύτηκαν όλους οι συγητές. Ναι, έκαναν ευρύτατη διαβούλευση, αλλά... Είναι η πρώτη φορά που είδαμε ένα σχέδιο έκθεση στην Επιτροπή. Και δεν νομίζω πως μπορούμε να πούμε πως υπάρχει συνένεση ακόμα. Για να διευκρινίσω αυτά που είπα προηγουμένως μετά από την παρέμβαση του Άντριου Ντάφ. Οι διαπραγματεύσεις, οι άτυπες διαπραγματεύσεις μεταξύ των συνεισηγητών και του Συμβουλίου θα αρχίσουν επίσημα μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Οπότε θα είναι η διαμορφωμένη θέση της Επιτροπής. Τότε θα έχουν την εντολή, οπότε περιμένουμε στο μεταξύ να μας ενημερώνουν για το πώς διαπραγματεύτηκαν το θέμα με το Συμβούλιο. Νομίζω ότι αυτή είναι η γραμμή συνένεση που έχει διαφάνει. Από αυτό το σημείο πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε εντό του έτου. Γι' αυτό και θα πρέπει να καταθέσουμε τι απολογίε όσο γίνεται πιο σύντομα. Ο Νταφ πάλι δεν συμφωνεί. Μα υπάρχουν αποκλήσεις, αλλά είναι ξεκάθαρες. Δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι αρκετά απλό. Έχει δίκιο ο Μέντες που λέει ότι οι διαπραγματεύσει είναι άτυπε μέχρι ότου να υπάρχει τελική ψηφοφορία τη Επιτροπή. Όμω αυτή η τελική ψήφο θα πρέπει να γίνει γρήγορα. Και αυτό προτείνω, να οριστεί η συζήτηση για τις 29.30 του μήνα. Και μέχρι τότε δεν θα υπάρχει επίσημη εντολή. Θα πρέπει να έχει κάποια ισχύ ενδεικτική η ψήφος. Εγώ δεν μπαίνω στην ουσία γιατί είμαι πρόεδρος, ε, αλλά κάποιες επιφυλάξεις έχω. Η πρωτοβουλία των πολιτών είναι πολύ σοβαρό θέμα. Για παράδειγμα, Να πούμε, την ε, δυνατότητα επιβεβαίωσης της ταυτότητας των πολιτών που την συνυπογράφουν, ε, να μπορεί να και στο κράτος ε, κάποιο δείγμα, να υπάρχουν προβλέψεις για τις ταυτότητες ή για τα διαβατήρια, κάπως να μπορούν να εντοπιστούν αυτοί που υπογράφουν, να αναγνωρίζονται, εν πάση περιπτώσει. Ε, τροπολογίες που θα αξιολογήσουν οι άτυποι διαπραγματευτές και που ε, μετά θα ψηφίσουμε μεγαλύτερη βεβαίωση. Εσείς σας είδα ότι διαφωνείτε, συνάδελφε Ντάφ. Ωστόσο πρέπει να αποφασίσουμε γι' αυτό. Εγώ προτείνω 15 του μηνό για την υποβολή των τροπολογιών και συζήτηση 20-29 του μηνό. Νταφ. Ναι. Εγώ ευχαρίστω να δεχτώ τι ε, προθεσμίε που είναι την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα. Πότε είναι 15. Σε 15 μέρες. Όχι. Τη Δευτέρα είναι 15. Τη Δευτέρα έχουμε 15. Δηλαδή νωρίτερα από ό,τι νόμιζα. Αλλά εντάξει. Θα δουλέψουμε το Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να βάλετε την προθεσμία στις 12 τα μεσάνυχτα τη Δευτέρα για να μας βοηθήσετε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν μπορώ να εγκρίνω αυτό το σχέδιο εντολής ως έχει τώρα. Also, ähm, ich bedanke mich. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Συμφωνώ ότι πρέπει να επιταχύνουμε προς την κατεύθυνση επίσημης εντολής και επομένως ψηφοφορίας στην Επιτροπή το δυνατόν σύντομότερο. Αυτό αναμένεται από εμάς άλλωστε και όντω θέλουμε να επιταχύνουμε. Συμφωνώ λοιπόν με την προθεσμία. Επισημαίνω μόνο το εξή, κάτι που είπα χθε ήδη στην συνάντηση των συντονιστών, ότι δηλαδή θεωρώ ότι και στις ανεπίσημες αλλά και στις επίσημες διαπραγματεύσεις θα πρέπει να συμπεριφθούν όλες οι πολιτικές ομάδες και όχι μόνο εκείνες οι οποίες έχουν ε, τους εισηγητές. Είναι σημαντικό το θέμα, ειδικά αυτός ο μηχανισμός να είναι να προκύψει μέσα από μια πολυφωνική συμμετοχή όλων των πολιτικών ομάδων. Αυτό νομίζω ότι αποτελεί μια δυνατότητα για το πώς μπορούμε αποτελεσματικά και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να οδηγηθούμε σε ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και με τα άλλα θεσμικά όργανα. Οπότε 15 λοιπόν, για τις τροπολογίες και 29 για τη συζήτηση. Δεν υπάρχει επίσημη εντολή. Υπάρχει δυνατότητα να συνεχιστούν οι σχέσεις αντεπισήμως και όταν θα έχουμε τελική έκθεση θα αποφασίσουμε καλύτερα για τη σύσταση της διαπραγματευτικής ομάδας. Συμφωνείτε? Έχουμε λίγα λεπτά, αλλά θέλω να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο Τερνέιρο και έπειτα στον κύριο Έρμπαντ του Συμβουλίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Καταρχήν να ευχαριστήσω για τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι στιγμής και ευχαριστώ τους εισηγητές για τη δουλειά που έκαναν, για τις διαβουλεύσεις που έγιναν. Είμαι αισιόδοξο ότι θα κάνουμε σημαντική πρόοδο να πιστήσω την προσοχή σε τρία σημεία, να μην επαναλάβω τα όσα έχουν ήδη υποθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις, να μην την προσοχή σε δύο-τρία σημεία, όπου υπάρχουν νέα στοιχεία ή που είναι τα πιο σημαντικά. Καταρχήν είναι αυτό το θέμα ανάμεσα στον έλεγχο της, ε, του παραδεκτού και την Επιτροπή των Πολιτών. Να διευκρινίσω ότι το κείμενο τώρα, όπως προτείνεται, λέει να εγκαταλείψουμε την ιδέα του να γίνεται ο έλεγχος ε, του παραδεκτού μετά από 300.000 υπογραφές και να γίνουν όλα εξ αρχής. Από... Ε, με τη διατύπωση που προτείνεται λοιπόν εδώ, στην ε, τροπολογία 27 νομίζω, είναι πρόοδος αυτό. Και αυτό συνδέεται στενά με το θέμα της Επιτροπής των Πολιτών, διότι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία με αυτόν τον τρόπο, αν από την αρχή έχουμε ένα είδος φίλτρου που μας επιτρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε γνήσια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία των πολιτών και ότι όχι κάποιος που ξαφνικά του ήρθε το πρωί ε, που ξύπνησε ξεκινά μια πρωτοβουλία και έχουμε να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Βλέπω τις δυσκολίες βέβαια το που μας ανέφερε ο κύριος Νταφ, αλλά είναι μια, μια σύνδεση ανάμεσα στα δύο. Πρέπει επίσης να σκεφτούμε αν κάποιος δεν μπορεί να βρει έξι ανθρώπους σε διάφορες χώρες για να στηρίξουν την ιδέα, τότε πώς μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος να ισχυριστεί ότι θα συλλέξει ένα εκατομμύριο υπογραφές από διάφορες χώρες. Χρονικός περιορισμός. χρονικός περιορισμός. Ένα άλλο ο περιορισμός που είναι η ακρόαση. Όταν δείτε τη 40-45 τροπολογία, θα δείτε εκεί ότι υπάρχουν δύο ακροάσεις. Μία πρώτη ακρόαση, όπου λέει ότι η Κομισιόν θα δεχτεί τους διοργανωτές στο κατάλληλο επίπεδο, ώστε να τους επιτρέψει να εξηγήσουν τα θέματα που θίγει η πρωτοβουλία. Αυτή είναι η πρώτη δυνατότητα ακρόασης, δηλαδή μια είναι μόνο μια γραπτή ε, διαδικασία ανάμεσα στον οργανωτή και την Κομισιόν. Θα υπάρξει μια διαδικασία ακροματική, ας πούμε έτσι. Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Εκεί που είναι το πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που το σχέδιο καθιστά αυτή την ακροματική διαδικασία υποχρεωτική που θα πρέπει να διοργανώνεται από την Επιτροπή, πιστεύουμε ότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δημιουργηθούν πολιτικές δυσκολίες, γιατί η Κομισιόν είναι ο παραλήπτης της πρωτοβουλίας, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι ουδέτερη, ότι είναι η προκατελημένη όταν οργανώνει μια τέτοια κρόαση. Άρα λοιπόν είμαστε πεπισμένοι ότι αν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, να επιβάλλουμε δηλαδή μια δημόσια κρόαση εκτός από την ε, ε, πραγματική διαδικασία, πιστεύουμε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διοργανώσει την ε, ακρόαση. Εδώ ο διοργανωτής θα αισθάνεται πιο, πιο άνετα και η Κομισιόν θα την προσωπεύεται, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην αρμόδια επιτροπή, στην Επιτροπή Αναφορών. Κύριε Χέρεμπο, εκπρόσωπος ε, του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά λακωνικός. Εκ μέρους της Βελγικής Προεδρίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές για το σχέδιο έκθεσης που κάνει ένα ακόμη βήμα πρόοδου προκειμένου να εγκριθεί το συντομότερο δυνατό κανονισμός ή ε, δυνατό και στα πλαίσια της πρώτης ε, επαιτίου εφαρμογής της συνθήκης Λισαβόνας. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες για να βρούμε συμβαστικές λύσεις για όλα τα θεμελιώδη ζητήματα και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να σας ικανοποιήσουμε σε πολλά σημεία. Οι μέχρι στιγμή συζητήσει πάντω έδειξαν ότι υπάρχουν ορισμένα σημεία που είναι ευαίσθητα για το Συμβούλιο. Οπότε εκεί εμείς θα ζητήσουμε την κατανόησή σα και πνεύμα συνεργασία. Ένα από αυτά τα θέματα αναφέρθηκε από πολλούς και αφορά την εξακρίβωση των υπογραφών. Το Συμβούλιο συμφωνεί απόλυτα με το στόχο σας να γίνει ο κανονισμός όσο πιο απλός και φιλικός προς τον πολίτη γίνεται. Όπως όμως επισήμαναν μερικοί, ένα, ένας μηχανισμός για να είναι αξιόπιστος προϋποθέτει την ε, εξακρίβωση των υπογραφών των συμμετεχόντων στην πρωτοβουλία αυτών των πολιτών. Γιατί αναφέρθηκε ένα μηχανισμό που θα είναι φιλικό προ το χρήστη, αλλά θα πρέπει να είναι φιλικό και προ τα κράτη-μέλη. Και αυτή η φράση, φιλικό προ τα κράτη-μέλη, νομίζω ότι θα έχει λαμπρό μέρο στο Συμβούλιο. Ζητώ λοιπόν την κατανόησή σα. Κάθε χώρα θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα μέσα και τους μηχανισμούς που έχει στη διάθεσή του, στη διάθεσή της, ανάλογα με, τη με την ένομη τάξη του και τη διαδικασίες που εφαρμόζει προκειμένου να προβεί στην εξακρίβωση των υπογραφών. Αυτό είναι το πιο ευαίσθητο θέμα και κανένα δύο άλλα σημεία. Το θέμα της ελάχιστης ηλικία και η περίοδος εφαρμογής για το κανονισμό. Πάντως προσβλέπω στη συνέχιση της καρποφόρας συνεργασίας με το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάφορες συζητήσεις που θα γίνουν σε επίσημο αλλά και σε άτυπο επίπεδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους διερμηνείς που εξακολουθούν να είναι παρόντες και θα παραμείνουν ε, για ακόμα 5-6 λεπτά κατόπιν δικού μου γενικού αιτήματος ε, γιατί πρέπει να δώσουμε το λόγο και στους δύο κύριος Λαμασούρη, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους διερμηνείς να πω δύο-τρία πράγματα. Θα ήθελα καταρχήν... Θα ήθελα καταρχήν να καθησυχάσω τον Άντριου Νταφ για το θέμα της Επιτροπής των Οργανωτών. Διαλέξαμε το 7 γιατί το 7 είναι ιερός αριθμός, συμβολικός αριθμός. Είχαμε τα 7 ουράνια σώματα που βλέπουμε πριν ε, θα έπρεπε να δούμε στον ουρανό πριν την ε, εφεύρεση του τηλεσκοπίου στην αρχαία Ελλάδα για παράδειγμα. Και υπάρχει κάποια συνάφεια στο τέλος μεταξύ του αριθμού των ε, συντακτών που συμμετέχουν στην Επιτροπή Οργάνωσης και του αριθμού των χωρών. αν έχουμε 5, 10 ή 7 χώρες, είναι λογικό να ζητούμε έναν εκπρόσωπο ανά χώρα. Και μάλιστα τη σήμερα ημέρα που έχουμε το διαδίκτυο, ένας πολίτης δεν μπορεί να βρει 6-7 πολίτες από άλλες χώρες. Πώς είναι δυνατόν να μπορεί ο ίδιος να συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο υπογραφές μέσα σε τρία χρόνια. Όπως και εσείς συμμετέχω στο facebook και έχω καταλήξει μέχρι και να, συντάκ, να, να γράφω γαλλικά χαϊκού κατά το γιαπωνέζικο πρότυπο για να συνομιλήσω με τον πρόεδρο Βανεροπόη. Κάθε φορά που συντάσσω ένα χαϊκού, αμέσως έχω 50 ε, αντιδράσεις από διάφορες χώρες. Βλέπετε, είναι η εποχή του ίντερνετ, η επικοινωνία είναι ελεύθερη, ε, εύκολη. Σε ό,τι αφορά την τροποποίηση, την αναθεώρηση των συνθήκων, εκεί δεσμευόμαστε από τις συνθήκες. Αν πούμε στον κανονισμό ότι μια πρωτοβουλία των πολιτών μπορεί να ακυρώσει συνθήκη, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα ακυρώσει τον ίδιο τον κανονισμό. Όπως είπε και ο κύριος Τσαρκόφσκι, προβλέπουμε ότι οι πολίτες... Ε, μάλλον υιοθετήσαμε μια διατύπωση που είναι σχετικά χαλαρή. Δεν έχουμε συγκεκριμένη μνήμα των άρθρων. Λέμε κάποια σχέση με τις διατάξεις της συνθήκης. Αυτή η γενική διάταξη αφήνει ένα περιθώριο λιγμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα κληρύνει το παραδεκτό για περιπτώσεις που βρισκόμαστε στα όρια των συνθήκων. Αλλά δεν μπορούμε επίσημα να δεχτούμε μια πρόταση, μια πρωτοβουλία για την ε, αναθεώρηση της συνθήκης. Σε ό,τι αφορά την εξακρίβωση ταυτότητας. Και εκεί υπάρχει διάσταση απόψεων. Υπάρχει μια συμβαστική πρόταση που υποβάλαμε προς τα κράτη-μέλη. Γιατί για τα κράτη-μέλη είναι δύσκολο αυτό το θέμα. Προτείνουμε λοιπόν στον κανονισμό να μην υπάρχει υποχρέωση χορήγησης αδελτίου ταυτότητας, αλλά υποχρέωση του υπογράφοντος να δηλώσει υπεύθυνα ποια ή τι είδους ε, ε, επίσημο έγγραφο μπορεί να πιστοποιήσει την ταυτότητά του. Δεν μιλούμε για αδελτίο ταυτότητας, μπορεί να είναι ε, ε, βιβλιάριο υγείας ή κοινωνικής ασφάλισης, άδεια οδήγησης και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αυτή είναι μια συμβαστική λύση που θα μας επιτρέψει να ξεφύγουμε από αυτό το διέξοδο. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ. Για τους υπογράφοντες. Φυσικά μόνο Ευρωπαίοι πολίτες μπορεί να είναι οι υπογράφοντες. Τώρα, ένας Πολωνός υπήκος μπορεί να κατοικεί στην Πολωνία. Δεν ξέρω αν κατοικεί στο Βέλγιο, αν θα το χαρακτηρίσουμε Βέλγιο ή Πολωνό. Αυτό μπορούμε να το ε, ρυθμίσουμε. Πάντως, ένας ε, Ευρωπαίος πολίτης που διαμένει στις Ινδίες, στις Ινδίες, ε, στη Σιβηρία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω αν μπορεί να συμμετέχει στην πρωτοβουλία των πολιτών. Μάλλον ναι, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε στην πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών να συμμετέχει ένας υπήκος τρίτης χώρας η κυρία Κοράτσα Μπίλτ είπε ότι θα πρέπει να αποκλείσουμε τους ε, αιρετούς ε, εκπροσώπους από τη ε, δυνατότητα συμμετοχής σε μια επιτροπή διοργάνωσης. Τι, να πούμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτών, δηλαδή οι αιρετοί και οι υπόλοιποι και δίνουμε το δικαίωμα σε όλους τους υπόλοιπους αλλά όχι στους αιρετούς γιατί έχουν δικαιώματα από άλλες πηγές. Εγώ διαφωνώ. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη των συνεισηγητών. Πάντως θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να γίνει διάκριση μεταξύ των βουλευτών και των άλλων. Αν απαγορεύσουμε σε ένα δημοτικό σύμβουλο ε, ενός μικρού χωριού, μικρής ε, πόλης να συμμετέχει, δεν ξέρω αν έχει νόημα. Όχι ότι απαγορεύουμε τη συμμετοχή σε μια επιτροπή διοργάνωση, αλλά να πούμε, αν ε, εγκρίνουμε το ελάχιστο όριο των 7, δεν ε, συνυπολογίζουμε στους 7 τους βουλευτές. Αυτό δεν τους εμποδίζει να συμμετέχουν, δεν εμποδίζει τους βουλευτές να συμμετέχουν στην ε, Επιτροπή Οργάνωση, γιατί 7 είναι το ελάχιστο όριο. Δεν ε, προβλέπουμε ανώτατο όριο. Απλώς δεν συμμετέχει, δεν συνυπολογίζεται ο βουλευτής στο ελάχιστο όριο των 7. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια πιθανή λύση. Τέλος, ε, το πρόβλημα που επισήμανε ο κύριος Γκερέρο. Δεν ξέρω πραγματικά τι να κάνουμε κύριε Γκερέρο για μια πρόσφατη νομοθεσία που μετά από μια χρονοβόρα διαδικασία συζήτηση, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Εγκρίνεται λοιπόν και μετά από λίγο συγκεντρώνεται πρωτοβουλία των πολιτών για να καταρρύψει αυτή τη νομοθεσία. Το συζητήσαμε αυτό το θέμα. Είναι ανοιχτό ερώτημα. Okay, I know our uh, να ξέρω ότι οι διερμηνεί μα είναι πολύτιμοι. Θέλω να του ευχαριστήσω για... και ευχαριστώ όλους σας για την συζήτηση. Ε, ελπίζω να μα βοηθήσετε με καλέ τροπολογίε να καταστήσω φές για όλου ότι όλοι μας προσπαθούμε να έχουμε καλή συνένεση και εγώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω να διατηρήσουμε αυτή τη συνένεση. Ευχαριστώ όλους ιδιαίτερος ε, την Γραμματεία, την Πάολα, Τάμας ε, και όλους που μπόρεσαν να μας βοηθήσουν ε, και τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ας προσέξουμε λοιπόν να κάνουμε καλή δουλειά. Ευχαριστώ και τον πρόεδρό μα που βοήθησε για αυτή τη διαδικασία, αλλά και ευχαριστώ και την κοινωνία των πολιτών που συμμετέχει ε, στην ε, δουλειά αυτή. Ας συνεχίσουμε και σκαταστήσουμε σαφέ ότι ελπίζω ότι θα έχουμε καλέ τροπολογισμέ μέχρι 20. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά από αυτή την πολύ σκληρή συνεδρίαση, δύο συμπεράσματα. Πρώτον, ε, επιβεβαιώσαμε τη δέσμευση να τελειώσουμε μέσα στον χρόνο αυτό. Δεύτερον, διαπιστώσαμε συνένεση που δεν αφορά όλα τα πάντα, αλλά την ουσία ότι υπάρχουν ε, λεπτομέρειες τις οποίες διαφορούμε και θα προσπαθήσουμε να τις λιάνουμε με τη βοήθεια των εισηγητών και με τη συζήτηση που θα κάνουμε στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ όλους. Τι πρέπει ακόμα να κάνω. Α, ναι, ναι, πολύ σημαντικό. Είχε ήδη αποφασιστεί και επιβεβαιώνω ότι υποβολή τροπολογιών μέχρι τις 15 του μηνό στι 12 το μεσάνυχτα. Όχι, όχι, συλληπάμαι. Εγώ ζήτησα... Α, συγγνώμη, δεν το άκουσα, δεν το άκουσα. Ναι, ναι, είπαμε με, μεσάνυχτα, μέχρι τα μεσάνυχτα. Ωραία, τέλος συνεδρίασης.